Uh, so good afternoon, everybody. I think we'll make a start. We're slightly, um, we're slightly light on shadow rapporteurs. Καλησπέρα. Δεν έχουμε όλους ακόμη τους πιο δυσυγητές, αλλά έχουμε τον Denis Διώ, τον εισηγητή μας, που είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως έπρεπε να σε φέρουμε στα μπροστινά έδρανα, αλλά μάλλον τώρα είναι αργά. Έχουμε την κυρία Κόνιν Λάγκεν, που εκπροσωπεί τον κύριο Σουβάπ, κυρία Πέντεργκάστ απουσιάζει. Φαντάζομαι κάποιος θα εκπροσωπεί το, τους σοσιαλιστές. Εγώ θα αντικαταστήσω το Σκιώδη γιατί κύριο Μπιέλλαν. Και με ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσω για την πρώτη συζήτηση την κυρία Μανφρέντι από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη Εσωτερικών Αγοράς και Καταναλωτών. Καλωσορίζω και εσάς και το επιτελείο σας και να σας υπενθυμίσω να καλωσορίσουμε φυσικά και το κοινό μας, τον κόσμο που μας παρακολουθεί με πολύ ενθουσιασμό για το θέμα αυτό από το διαδίκτυο στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίας της Επιτροπής και έχουμε και το δελτίο μας, το newsletter, το καινούριο που αν σας ενδιαφέρει μπορείτε άπαξ το μήνα να το λαμβάνετε, αναφέρει τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας. Πρόκειται για μια έκθεση της πρωτοβουλίας που διακαώς επιθυμούσαν να συντάξουμε οι συντονιστές προκειμένου να ασχοληθούμε με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, παραπλανητική διαφήμιση και άλλα σημαντικά θέματα που εξετάζει ο κύριος Διόν και έχουμε και την αναθεώρηση της οδηγίας Επιτροπής των Εμπορικών Πρακτικών υπό το πρίσμα του καταναλωτή. Έχουμε ήδη λάβει το σχέδιο έκθεσης του Δινιστίου. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις και του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών. Mrs. Ruler, Mrs. Ruler has arrived just in time, so we have an almost complete suite of shadows, but no one from the S&D yet. Έφτασε η κυρία Ρούλε στο μεταξύ. Έχουμε σχεδόν απαρτία σκιωδών εισηγητών. κυρία Στάιλερ, αν θέλετε να παίξετε το ρόλο κάποιου σκιωδού εισηγητού, είστε ευπρόσδεκτοι. Ντένις, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Να ξεκινήσω με μία συγκεκριμένη περίπτωση που υπέπεσε στην προσοχή μου μέσω του εστιακού σημείου, του εθνικού εστιακού σημείου κατά της απάτης. Υπάρχει μια εταιρεία, όμιλος εταιρεών ε, που λέγεται Business Group. Ακούστηκαν διάφορα παράπονα από εταιρείε που υπέπεσαν θύματα αυτής της πρακτικής της πρώτης εταιρεία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν. Οι εταιρείε θύματα ζήτησαν να ελεγχθούν τα στοιχεία της, του οδηγού της business της άλλης εταιρείας, της πρώτης εταιρείας. Ως ε, Ευρωβουλευτής ε, συχνά μου ζητάνε να ελέγξω αν τα στοιχεία σε ένα μητρό είναι σωστά. Και πάντα απαντάω ότι είναι ή δεν είναι σωστά. Αυτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί εντολή να γραφτούν σε αυτόν τον οδικό. Τα, στοιχεία ήταν σωστά, αλλά μέσω ε, μικρών λεπτομεριών ε, υποχρέωναν χωρίς να καταλάβουν οι εταιρείε, επειδή βάζαν τα στοιχεία τους απλώς, ότι γινόταν μέλη πληρώνοντας 75 ευρώ το χρόνο ε, ήταν κάτι στα ψηλά αυτό που γραφόταν, ότι πραγματικά ε, επρόκειτο περί σύμβασης. Και αυτά τα λεφτά πήγαιναν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στις κάτω χώρες. Και από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό, τα λεφτά που έφευγαν πήγαιναν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία. Σε μορφή ρευστού. Οι δικαιούχοι ήταν άλλες εταιρείε με λογαριασμού στο εξωτερικό. Υπάρχει μια διεθνοποίηση αυτών των εταιρείων και αυτός ο όμιλος των εταιρείων που ήταν πίσω από αυτόν τον οδηγό Eurobusiness είχε ένα call center, ένα κέντρο κλήσεων στη Ρουμανία. Ε, λεφτά πήγαιναν και σε εργαζόμενες σε αυτό το κέντρο. Το πράγμα περιπλοκόταν. Οι αρχές εφαρμογής του νόμου είχαν δυσκολίες. Ε, καταρχάς τέτοιου εγκλήματα είναι δύσκολο να ανοιχνευτούν και περιπλέκονται ακόμα περισσότερο γιατί ε, τα θύματα είναι από όλες τις χώρες και οι επιχειρήσεις επίσης είναι εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες, άρα άσε αυτή την ιστορία, ας μην την ψάξουμε, ε, είναι πολύ δαπανηρή, χρονοβόρα κτλ. Όταν, υπάρχει, όταν εμπλέκονται κρατημέλη, η περιπλοκότητα του πράγματος αυξάνεται. Αλλά αυτές οι τάσεις είναι πολλές και μπορούμε να κάνουμε πολλά σε αυτόν τον τομέα για να βελτιώσουμε το, τις επιδόσεις των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και τη συνεργασία τους. Δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι σημαντικό οικονομικά για τη χώρα. Τα νούμερα για την Ολλανδία είναι 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που χάνουν οι εταιρείε λόγω αυτών των πρακτικών. Τα μεμονωμένα ποσά είναι πολύ μικρά. Μόνο να τα προσθέσει όλα μαζί έχουν σημασία. Ε, σε τέτοιες εποχές όταν ας πούμε αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε εγκληματίες ε, είναι μεγάλη σπατάλη. Τώρα, πολλαπλασιάστε αυτό το νούμερο ε, επί χ για την Ευρώπη, άρα μιλάμε για δις. Δεν ξέρω πόσα, γιατί δεν είναι καταχωρημένα, αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά, συνολικά, όχι μεμονωμένα επαναλαμβάνω. Αυτό που προτείνω στην έκθεση είναι καταρχάς πρόληψη, διάφορα μέτρα που εντάσσεται στον τομέα τη πρόληψη, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται γι' αυτό εθνικά σημεία επαφή για κάθε κράτο. Έχουμε εμεί στην Ολλανδία ένα τέτοιο εθνικό σημείο επαφή. Είναι πολύ σημαντικό για του ε, επιχειρηματίε. που μερικέ φορέ ε, τραυματίζονται από όλε αυτέ τι ε, εμπειρίε. Μπορεί να μην θεωρηθεί, α πούμε, καλό επιχειρηματία. Δεν κατάλαβε ότι έπρεπε για κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβε ότι ήταν εγκληματική δραστηριότητα, αλλά αν υπάρχει ένα εθνικό σημείο επαφή, μπορεί να βοηθήσει. Εγώ πήγα σε αυτόν τον άνθρωπο και ένα από τα τηλεφωνήματα αυτά, μία από τις τηλεφωνικές κλήσεις, α, είχε καταγράψει ένας επιχειρηματίας, του τηλεφώνησε κλαίγοντας και του είπε ότι αισθάνθηκε και ταπεινωμένος αλλά και φοβισμένος πια από την ιστορία. Και το εστιακό σημείο θα μπορούσε να του δώσει όχι μόνο ε, συμβουλέ. Η βασική συμβουλή είναι μην πληρώνει. Μην πληρώνει, μην πληρώνει. Αυτή είναι η βασική συμβουλή. Αλλά πέραν αυτού καταγράφει και τι συνέβη και συσσωρεύει και τα δεδομένα που βοηθάει έτσι τις ε, ε, αρχές εφαρμογής του νόμου για να καταλάβουν δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο σημείο, αλλά είναι ένα μοντέλο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό Επίσης, ε, και νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Γιατί πρέπει να συνεργαστεί κανείς, οι εθνικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν με τις οργανώσεις των εργοδοτών. Υπάρχει η πραγματογνωμοσία από τη μεριά τους και στην Ολλανδία ε, λειτουργήσε αυτό και κάνω σύσταση στα άλλα κράτη-μέλη να το κάνουν, να το ψάξουν. Βεβαίως χρειαζόμαστε και ένα μαύρο κατάλογο ε, αυτών των ε, εταιριών που κάνουν τέτοιες ε, πρακτικές απάτης και ποιες είναι οι πρακτικές όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρείες, ταχυδρομεία, εταιρείε ίσπραξης κτλ. που υποβοηθούν αυτή την απάτη. Γιατί όλοι παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να τους αναγνωρίσουμε, να ξέρουμε ποιοι είναι και να σταματήσουμε, να τους σταματήσουμε, να μην τους επιτρέπουμε να είναι του προβλήματος, αλλά και η εφαρμογή του νόμου. Γενικά οι αρχές έρευνας, διερεύνησης, γενικά είναι απρόθυμες να ασχοληθούν γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά και αν δεν κάνεις τίποτα, ποτέ θα γίνει προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο. Δεν κάνει κανένα τίποτα, εν Γι' αυτό μια κάποια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν ε, ίσως θα ήταν καλό, ίσως κατευθυντηρίες γραμμές από την Κομισιόν. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αλλιώς ποτέ δεν πρέπει να γίνει προτεραιότητα αυτό το θέμα. Φυσικά χρειαζόμαστε και κυρώσει. Θέλουμε να τιμωρήσουμε δια νόμου αυτές τις πρακτικές. Είναι μερικές φορές δύσκολο να οι διοκτικές αρχές να μπορέσουν να βρουν αναφορές στα ίδια πατών σαπάτες ή σε παρόμοιες ε, απάτες που να περιγράφουν πραγματικά την ε, πραγματικότητα. Σε ορισμένε χώρες, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, υπάρχει ειδική νομοθεσία για τέτοιες ε, πρακτικές, για τέτοια αδικήματα και έτσι οι διοκτικές αρχές διευκολύνονται για να προβούν σε δράση. Η καταχώρηση των εταιριών είναι πολύ σημαντικό και οι εταιρείε με αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές θα πρέπει να εντοπίζονται αν είναι ύποπτες, ε, αν είναι ύποπτη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο αυτό σε αρχικό φας, ε, στάδιο. Ε, επίσης, οι εταιρείε ίσπραξης παίζουν το ρόλο τους και θα πρέπει να τις ελέγχουμε καλύτερα από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών ε, λείπει. Επίσης, υπάρχει ένα μικρό κεφάλαιο στην έκθεση για τη διεθνή συνεργασία, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάει αυτή η ιστορία στα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπάρχουν διεθνείς πρωτοβουλίες και ιδίω στην έκθεση αναφέρεται μια ομάδα εργασία που ασχολείται με τις πρακτικές marketing. Είναι μια άτυπη ομάδα, αλλά συνεργάζεται πολύ καλά. Φερρυπίν έχει σχέσεις με επιχειρήσεις ή με ιονή επιχειρήση στην Νιγηρία αυτή η ιστορία και δεν μπορείς να επιλύσεις τέτοια προβλήματα μόνος σου. Ε, επίσης, η συνεργασία με τις είναι πολύ σημαντική. Δεν μου μείνει και καθόλου χώρος για να πω οτιδήποτε για τη συγκριτική διαφήμιση, που είναι και αυτό το τμήμα της ανακοίνωσης της Κομισιόν, όπου βασιζόμαστε, ως προτεραιότητα θα έλεγα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την έκθεσή μου, που είναι λιγάκι μακρύτερη, μακροσκελέστερη από ό,τι συνήθως, λόγω των προβλημάτων που σας προανέφερα. Φυσικά, με, για τις τροπολογίες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε θέλει να ρυθμίσει και να αναφερθεί σε θέματα που αφορούν τη συγκριτική διαφήμιση μέσω τροπολογιών, κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ αν το κάνουν άλλοι. Τώρα για το φωνοδιάγραμμα και ας ε, επαληθεύσει η γραμματεία ότι λέω τα σωστά πράγματα. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, ε τροπολογίες είναι 18 Ιουνίου ε, μεσημέρι, 5 Σεπτεμβρίου θα τις εξετάσω μετά το καλοκαίρι δηλαδή. Μετά τις, τις συμβαστικές 25 Σεπτέμβρη, 26 Σεπτέμβρη ψηφοφορία και 2 Οκτωβρίου ή στη, στη δεύτερη ολομέλεια μάλλον του Οκτωβρίου θα υιοθετήσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Στις 8 ε, και 9 Ιουλίου θα κοιτάξουμε για ε, πρώτη φορά τις ε, τροπολογίες. Αλλά νομίζω έτσι καλώ πω πως συνεργάζεστε στενά με τους κοιόδης εισηγητές, οπότε μπορούμε να βρούμε κάποιο σημείο να τις εξετάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένις. Μας τα εξήγησες πολύ καλά. Υπάρχουν πάρα πολλέ συστάσει στην έκθεσή σου. Φυσικά, όπω συμβαίνει με κάθε εκθέση ε, ιδιαίτερη πρωτοβουλία, ο εισηγητή πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομο και περιεκτικός. Και δυστυχώ δεν έχουμε την ε, ευκαιρία λοιπόν να επεκταθούμε και να εμπλουτίσουμε την έκθεση, αλλά ο ρόλο των σχεδόν εισηγητών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν πάρα πολλά να συνεισφέρουν. Έχουμε πάρα πολλέ τροπολογίε, οι οποίε, ε, για παράδειγμα, ψηφίστηκαν σήμερα στην έκθεση του κυρίου Φόξ, οι οποίε δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενε. Όπω και να έχει όμω, α ακούσουμε καταρχά την ε, κυρία Κόλλιν Λάγκεν εκ μέρου του κυρίου Σφαμπ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Σφάμπ, ο οποίο δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να παρουσιάσω ορισμένα σημεία εκ μέρου του. Καταρχάς ευχαριστή πάρα πολύ εσάς, κύριε Ντεγιόγκ, για την έκθεση. Ο κύριο Σφάμπ σήμερα θα ήθελε να επικεντρωθεί σε δύο σημεία και να κάνει κάποιες σύντομε παρατηρήσεις για τις ε, τροπολογίες. Πιστεύω πως μπορούμε να το συζητήσουμε και στα και τα δύο σημαντικά σημεία αναφέρθηκαν ήδη, η μαύρη λίστα για τις ε, παραπλανητικές επιχειρήσεις και μια πρόταση για περαιτέρω ενίσχυση της ε, δομής και του συντονισμού του τοπισμού. Ο κύριος ε, Σβάμπ διατυπώνει τις σκέψεις του και τις αμφιβολίες του για το πόσο καλά θα λειτουργήσει αυτό, διότι δεν είναι ακόμα σαφές Ποιε από αυτές τις επιχειρήσεις θα μπουν σε αυτή τη μαύρη λίστα, πώς θα γίνεται η διαδικασία λήψη αποφάσεων και πώς θα γίνεται όλο αυτό. Πολλές φορές αυτές οι εταιρείε έχουν, ε, αλλάζουν την έδρα τους από το ένα, μέρος, από το ένα μέλος κράτος στο άλλο έτσι ώστε να αποφύγουν την ε, δίωξη. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σβά ε, πιστεύει πως καλύτερα θα ήταν να υπήρχε μια ε, πανευρωπαϊκή εμβέλεια σε μαύρη λίστα για αυτές τις ε, εταιρείε. Τώρα, όσον αφορά τον συντονισμό και την διοικητική δομή, η δημιουργία μιας εθνικής τράπεζας δεδομένων που έχει προταθεί είναι κάτι το οποίο είναι όχι και τόσο οικονομικά εφικτό, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στα μέσα μιας οικονομικής κρίσης. Πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε το κόστος να μην απομιστεί μόνο από ένα κράτος μέλος, αλλά να μοιραστεί. Ο κύριος Σφάμπε τονίζει ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες εμβάθυνσης και ενίσχυσης με τις δικές του τροπολογίες της υπάρχουσας δομής. Και αυτό είναι κάτι που έχει συζητήσει και στη... με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λάγεν. Παρακαλώ, θα θέλατε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική έκθεση και πραγματικά και στη Σκωτία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτές τις αθέμητε πρακτικέ και πραγματικά αγγίξατε τα ευαίσθητα σημεία ε, με την έκθεσή σας διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι αισθάνονται πως τους έχουν εξαπατήσει και μάλιστα έχουμε και λέξη που προσδιορίζει αυτούς τους απαταιώνες. Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα. Ο κόσμος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει επίσημες επιστολές από δικηγόρους. Γι' αυτό και χρειάζεται να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρήκα την έκθεσή σας πάρα πολύ χρήσιμη επίση, γιατί συμπεριλαμβάνονται και οι πρακτικέ των άλλων κρατών μέλων. Τι γίνεται λοιπόν εκεί. Και πραγματικά νομίζω πω αυτή η μαύρη λίστα που χρησιμοποιούν εταιρεών είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που δεν έχω καταλάβει καλά είναι τι γίνεται με τους επιμέρους κανόνες και τη μεταφορά των εταιριών αυτών από κράτος σε κράτος. Δεν έχω καταλάβει ακόμα εσείς πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε την πρακτική αυτή, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να πω ότι στηρίζω την έκθεσή σας. Είναι κάτι αναγκαίο, είναι κάτι που μας λείπει. Και πραγματικά να πω ότι μας ασκήθηκε πίεση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στην Επιτροπή Αναφορών είχαν ε, παραπεμφθεί τέτοια θέματα πάρα πολύ συχνά και πραγματικά μας κατηγορούσαν ότι δεν κάνουμε τίποτα και πρέπει να κάνουμε κάτι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι ιδιαίτερα εν ώψη των ευρωεκλογών του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ που μας μάθατε και καινούργια πράγματα. Κύριε Ρόσφορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Ντε για το έργο αυτό που ε, φυσικά θα τύχει και της δικής μας υποστήριξης και συνδρομής και θα έλεγα ε, ότι μερικοί ευρωβουλευτές ε, αυτοπαγιδεύθηκαν σε τέτοιου είδους ε, πρακτικές και γι' αυτό ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το θέμα που προβληματίζει και ταλανίζει δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα είναι εύκολη η συνένεση για την έκθεση αυτή σε θέματα όπως ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με καλύτερη ανταλλαγή των πληροφοριών και επίσης ε, ε, περιμένουμε την υπομονησία τη προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που υποσχέθηκε ότι στα μέσα του 2013 θα υποβάλει εξονυχιστική ανάλυση της κατάστασης προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Και το θέμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες επίσης είναι σημαντικό και εσείς μόνο σας με το παράδειγμα που μας δώσετε κύριε De Jong. μας είπατε ότι πρόκειται για δίκτυα που παραπέμπουν από χώρα σε χώρα, είναι και μερικές φορές εξωτερικά της Ένωσης, οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς έγκαιρες προειδοποίησης, ώστε να είναι άμεση αντίδραση και αποτελεσματική και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτό των σύνορων τη. Τώρα, ένα άλλο σημείο για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί μερικά προανέφεραν οι συνάδελφοι, ε, είναι ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της μαύρης λίστας των ε, απατηλών ή παραπλανητικών πρακτικών. Γιατί είναι γνωστές πια οι πρακτικές και καλό θα ήταν ε, να, περιγραφούν και σε, έναν, σε μια μαύρη λίστα. Και ίσως η μαύρη λίστα των πρακτικών θα μπορούσε να συνοδευτεί, να τη διαδεχθεί μια μαύρη λίστα των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω βέβαια θα πρέπει να στιγματίσουμε τις επιχειρήσεις ε, μετά τις πρακτικές, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι ειδικευμένε σε τέτοιου είδους απάτες και μερικές τέτοιες πρακτικές από μόνες τους ε, δεν είναι θέμα, δεν ανήκουν στην παιδεία της ε, εταιρείας, αλλά λόγω κάποιων αδυναμιών στη διαχείριση δημιουργήθηκαν τέτοιε ε, απατηλές πρακτικέ ω ε, παρενέργεια. Πάντως, ε, σίγουρα θα πρέπει να αποκλείσουμε τέτοιε εταιρείε που μετέρχονται απατηλών πρακτικών από του διαγωνισμού δημοσίων προμηθειών. Αλλά ίσω δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ βιαστικοί. γι' αυτό να ξανασκεφτούμε την παραγράφο 7, εκεί που μιλάμε για συνυπευθυνότητα των τραπεζών, ταχυδρομείων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Το ταχυδρομείο, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν πρέπει να, ελέγχει το περιεχόμενο των ε, επιστολών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο να αναλάβει τέτοια ευθύνη το ταχυδρομείο, να ελέγχει το περιεχόμενο αυτών που στέλνει. Επίσης υπάρχει και το θέμα, όπως είπατε και εσείς κύριε De Jong, στο σχέδιο της έκθεσής σας, το κατά πόσο θα πρέπει να επεκτείνουμε την ε, οδηγεί αυτή από τις, ε, από τις σχέσεις επιχειρήσεων καταναλωτών, σχέσεις επιχειρήσεων μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η, με, με, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή στι ε, σχέσει μεταξύ των επιχειρήσεων και στη χρήση τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων. B2B, όπω λέμε. Κάτι τέτοιο έχει γίνει ήδη στη Γαλλία. Οπότε, αν δημιουργηθεί μεταξύ μας συμφωνία σύντομα για να διευρύνουμε την οδηγία από σχέσεις επιχειρήσεων καταναλωτών και σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί όχι, να το σκεφτούμε. Ε, πολλά δε μάλλον που περιμένουμε και μία έκθεση που αφορά την αξιολόγηση της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Οπότε ούτως ή άλλως θα ασχοληθούμε με αυτή την οδηγία που διέπει τις σχέση επιχειρήσεων καταναλωτών. Ας περιμένουμε λίγο λοιπόν πριν να σπεύσουμε να περιλάβουμε στο δικό μας κείμενο αυτή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Και επίσης στην παράγραφο 16 της έκθεσής σας μιλάτε για την πιθανή χρήση των συλλογικών αγωγών. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ κατά τέτοιων συλλογικών μέσων προσφυγή, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων και εντό τη επιτροπή αλλά και εντό κάποιων πολιτικών ομάδων. Τώρα, μια και περιμένουμε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα συλλογικά ένδικα μέσα, ας μην προτρέξουμε εμείς αναφέροντας κάτι τέτοιο στη δική σας έκθεση. Ας περιμένουμε την έκθεση πρωτοβουλίας της, ε, την πρόταση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συλλογικά ένδικα μέσα, τις συλλογικές αγωγές. Και επευκαιρία εκείνης πρόταση να το συζητήσουμε. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να περιλάβουμε και τις εμπορικές πρακτικές, τις καταχρηστικές ε, και στο πεδίο εφαρμογή της επερχόμενης πρώτης Επιτροπής για τα συλλογικά έδικα μέσα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεγιούγκ και για την έκθεσή σας και για την προθυμία και το διαλλακτικό σας πνεύμα. Γιατί υποσχεθήκατε ότι θα εξετάσετε πολύ επικοδομητικά και τις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Τενίστε Young. Πιστεύω ότι η έκθεσή του περιέχει μια πραγματικά καλή ε, ανάλυση και απαντά στα σημαντικά σημεία τα οποία τα θέτει στο προσκήνιο και όλα αντί για το περιθώριο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, εταιρείες οι οποίες ε, βρίσκονται καταχωρημένες στους ε, τηλεφωνικούς καταλόγους και τις ε, παραπλανητικές πρακτικές ε, που γίνονται εκεί. Τα, προβλήματα είναι πραγματικά υπακτά. Και πολλές φορές ε, δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη τα θύματα, διότι τα ποσά είναι μικρά, δεν είναι τόσο μεγάλα. Αλλά πραγματικά να πω ότι χαίρομαι, γιατί σε μία περίοδο που το πρόβλημα αυτό οξύνεται, πραγματικά αποφασίζουμε και ενδιαφερόμαστε για τους ε, πολίτες και αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα τους ωφελήσει. Δύσκολο όμως θέμα θεωρώ πως είναι οι λύσεις. Η καλή προετοιμασία των κρατών μελών είναι μεταξύ άλλων πολύ χρήσιμη και πολύ λογική και φυσικά η ανταλλαγή των πρακτικών είναι κάτι το σημαντικό και η συνεργασία με διεθνείς ε, ομάδες αντιμετώπισης. Ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση έχουμε εντοπίσει τα δύσκολα σημεία, ιδιαίτερα τα, ε, τις δυσκολίες ε, που αφορούν τις ε, δημόσιες, τους δημόσιους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις. Πιστεύω πως πραγματικά πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί, να το αναλύσουμε, να σκεφτούμε ποιες προτάσεις είναι εφικτές, τι μπορούμε να κάνουμε, από πού μπορούμε να αρχίσουμε να πιάσουμε το κουβάρι. Όταν συζητούσαμε την οδηγία για τις ε, αθέμητες πρακτικές, θυμάμαι ότι πάρα πολλοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να επεκταθεί το ε, από B σε B. Και φυσικά όσον αφορά τις συλλογικές προσφυγές γνωρίζω ότι αυτό είναι κάτι αρκετά αμφιλεγόμενο, όμως έχει καταστεί σαφέ ότι αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όταν τα ποσά τα οποία ε, παίρνουν εξαπατώντα τις επιχειρήσεις είναι μικρά και το κόστος μιας δίκης είναι πάρα πολύ υψηλό. Ελπίζω πραγματικά μαζί να βρούμε μια κοινή λύση. Όμως, ε, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θίξατε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που όλα και οξύνεται. Ε, ευχαριστώ. Ω και όλες θα μιλήσω τώρα, αλλά και ω άτομο που ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το θέμα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τι παραπλανητικέ εμπορικέ πρακτικέ, συμφωνώ με την κυρία Ρούλε. Είμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο πολύ καιρό και αυτό το θέμα πιθανής επέκτασης στη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων έχει ξανακουστεί, αλλά υπάρχει μεγάλη αντίθεση, αντίδραση από τα κράτη-μέλη. Ως βραχυπρόθεσμο, έτσι, βραχυπρόθεσμο μπάλωμα δεν νομίζω ότι είναι καλό. Αλλά για τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και για να το πω έτσι ήπια, ε, υπάρχει ασυνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης. Δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές ε, τα ίδια δικαιώματα και τα ίδια ένδικα μέσα στη διάθεσή τους, για να μην πω για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι σωστό αυτό. Και επίσης, όπως είπατε κι εσείς, οι πρακτικές παραπλανητικής διαφήμισης, αυτές μπορούν να αφορούν καταναλωτές, επιχειρήσεις και ο καθένας να τις κάνει ωραιότατα από μόνος του. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, αν εντοπίσουμε και ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχουμε αυτά τα παραπλανητικ... τους παραπλανητικούς οδηγούς επιχειρήσεων. Είναι απάτη πραγματική από λαμόγια πραγματικά και είναι ε, στα όρια της νομιμότητας, επίτηδες το κάνουν έτσι. Στην παράγραφο 8 του κειμένου σας πολύ σωστά λέτε ότι τα κράτη-μέλη ε, ήταν πολύ απρόθυμα να αναλάβουν και να ασχοληθούν περιπτώσεις παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ γιατί δεν, έχουν, δεν υπάρχουν και σαφείς αποδείξεις. συχνά ε, από τα ψηλά αυτά τα συμβόλαια, αυτό το mailing κτλ. περνάει σε μεγαλύτερους χαρακτήρες, ούτως ώστε να μην τους κατηγορήσει κανείς ε, για παραπλανητική πρακτική. Ε, τέτοιες, τέτοια αιτήματα μου φτάνουν και εμένα, γιατί ε, ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι αλλάζουν αυτές οι πρακτικές. Τώρα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αναγκάζει κάπου να καταχωρήσει το ΦΠΑ σε κάποια βάση δεδομένων, ε, χρησιμοποιούν αυτό το, το γεγονός και αλλάζουν τις πρακτικές απάτες. Δηλαδή δεν έχουμε πια τους κλασικούς αυτούς οδηγούς ε, εταιριών. όλα αυτά τα λέω πολύ προσεκτικά. Συμφωνώ με αυτά που η κυρία Λάγκεν εκ μέρου του κυρίου Σουβάμπ. Το πρόβλημα είναι ότι βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας αυτές οι πρακτικές. Το να προσπαθήσουμε επίσημα να τις βάλουμε σε μαύρη λίστα μπορεί να, δημιουργηθούν, να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να δίνουν παραδείγματα του τι δέχονται σε, όχι σαν μητρό, να μην το πούμε καν μητρό, κάπου τέλο πάντων, τόσο ώστε να ξέρουμε περί πρόκειται και να το βλέπουν και οι άλλοι επιχειρηματίε. Να έχουμε δηλαδή α, κάθε νέα υπηρεσία, οτιδήποτε σου προτείνουν τέτοιου τύπου που, είναι στα όρια της νομιμότητας, να κυκλοφορεί κάπου να ανακαταχωρημένη ας πούμε, ως πρακτική για να τη βλέπουν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες για να εξοικειώνονται. Γιατί η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε ό,τι αφορά τις απάτες. Είναι καλές αυτές οι ιδέες. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης και τις οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να τις ενθαρρύνουν να το κάνουν. Αν θεωρούν ότι υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια, να τα άρουμε. Ε, η κυρία ε, Στάιλερ είπε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Solvit για να παρακάψουμε το πρόβλημα. Ενημέρωση προς επιχειρήσεις είναι η λύση. Εγώ χρησιμοποίησα το δικό μου email πρόσφατα και παρατήρησα ότι έχω φτιάξει μια μικρή δική μου προσωπική βάση δεδομένων και στέλνω πληροφορίες σε διάφορους. Ε, με αυτόν τον τρόπο ειδοποιώ τον κόσμο. Στην τελευταία ειδοποίηση που έκανα έλαβα και πολλές απαντήσεις. Ε, ορισμένοι με ευχαρίστησαν που τους ενημέρωσα, που, μου, που τους επέσα την προσοχή κτλ. Είναι μια μικρή περιπέτεια αυτή. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να, να προωθήσουμε και να την συζητήσουμε αυτή την ιδέα με την, ή αυτές τις ιδέες πάμε, με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ε, για να έχουμε ιδέα για το πώς ασχολούνται, πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα επιχειρήσεις. Τώρα, για άλλες ιδέες που ακούστηκαν. Ορισμένες είναι επικίνδυνες γιατί μπορεί να είναι επιζήμιες και όχι υποφελεί. για τις δημόσιες προμήθειες. Αν κάποιος θεωρείται ότι έχει διωχθεί για παραπλανητική διαφήμιση, κυρία Ρούλε, σε εσάς στρέφομαι, γιατί τα ξέρετε αυτά. Τότε αποκλείεται από ένα διαγωνισμό, έτσι, μόνο και μόνο, γιατί έχει καταδικαστεί γιατί έχει γίνει δημόσια, ε, του είχε ασκηθεί δίωξη. Και αν έχει υπάρξει πρόβλημα με την φορολογία και τα λοιπά κάποιες επιχειρήσεις. Τώρα, για τις λογικές αγωγές. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις οργανώσεις των επιχειρήσεων να ασκούν τέτοιες αγωγές. Όπως είπε και ο Τόνι, ε, για, είναι πολύ σωστή η ιδέα της ε, ενημέρωσης, γιατί ακριβώς αυτές οι πρακτικές αλλάζουν πολύ γρήγορα και οι επιχειρήσεις, αυτές οι απατηλές ας πούμε, ε, μετακινούνται από μέρος σε μέρος. Τώρα, κάτι γενικότερο θέλω να πω για την ε, συμπεριφορά που είναι κατά του ανταγωνισμού ή που είναι αθέμητη ή στρεβλή. Να σας υπενθυμίσω, όταν συζητήσαμε την, τα δικαιώματα των χρηστών ε, στις καθολικές υπηρεσίες, πακέτο τηλεπικοινωνιών ήταν αυτό, συζητήσαμε το θέμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ε, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλο για να τα εφαρμόσουμε και για τις μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή κάτι, κάτι παρόμοιο. Και υπάρχει μια ρήτρα Τώρα τα μπέρδεψα όλα. Μιλάμε για το κείμενο, την οδηγία για τι καθολικέ υπηρεσίε, που υπάρχει μια διάταξη όπου οι ρυθμιστικέ εταιρείε των επικοινωνιών μπορούν, αν θέλουν, να επεκτείνουν κάποιε από τι διατάξει στι μικρέ επιχειρήσει. Θα κάνω μια έκθεση για την εφαρμογή αυτού του κειμένου στην Επιτροπή. Από ό,τι ξέρω, κανένα δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τέτοια πράγματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Απλώ θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά τα θέματα οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να δουν τι μπορούμε να κάνουμε ας πούμε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι μπορούν να κάνουν. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά. Δικά μου. Όλα τα άλλα όμως τα λέω ε, εκ μέρους του κυρίου Μπιέλαν. Αυτά από μένα. Θέλει κανένας άλλος να πει τίποτα. Ουδής. Ο κύριο Μανφρέντι. Η κυρία Μανφρέντι. Να απαντήσει σε όλα όσα της είπαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομε δηλώσει αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε έναν πανευρωπαϊκό, ε, μια πανευρωπαϊκή μελέτη αντικτύπου για το φαινόμενο αυτό θα συγκεντρώσουμε πολλά στοιχεία και ήδη έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη και πολύ φοβόμαστε ότι το ορατό σημείο είναι μόνο η κορυφή του παγόβανου. Φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις δεν τολμούν καν να παραπονεθούν ε, και να καταγγείλουν τις πολλές φορές που έγιναν θύματα τέτοιου είδους ε, αθέμητων και απατηλών εμπορικών πρακτικών. Το επισημάνατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτή το, τη μελέτη αντικτύπου που θα μας ε, παράσχει αδιάστα τεκμήρια για το έβρος του φαινομένου αυτού, κάτι που δικαιολογεί την επιτακτική ανάγκη άμεση ανάληψης δράσης. Και μάλιστα, όπως ήδη είπαμε στην περσινή μας ανακοίνωση, θα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ε, νομοθετική αναθεώρηση για τα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιδέα της ε, διεύρυνση όχι της προστασίας που παρέχουμε στους καταναλωτές ε, με την οδηγία κατά των πρακτικών και στις επιχειρήσεις, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ε, εξάγουμε από αυτήν την οδηγία για τις αθέμητες πρακτικές το απάβγασμα της προστασίας και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις παραπλανητικές πρακτικές marketing και στη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να το παρακάνουμε. Θέλουμε το απαραίτητο επίπεδο προστασίας Οπότε σίγουρα η οδηγία αυτή για την προστασία των καταναλωτών στι σχέσει με τι επιχειρήσει θα είναι το πρότυπο, το υπόδειγμα για να δράσουμε, αλλά προ το παρόν είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα ήταν σκόπιμο ούτε σωστό να το παρακάνουμε και τι απαιτήσει για διπλή πληροφόρηση που προβλέπει η οδηγία αυτή ε, για τι σχέσει καταναλωτή επιχείρηση να το επεκτείνουμε και στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρησεων σχεσει σχέση B2B που λέμε τι είναι προς το παρόν η, και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από στοιχεία που συγκέντρωσε. Τώρα, μία μικρή δήλωση, μία σύντομη δήλωση για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την διασυνοριακή συνεργασία και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το κατά πόσο θα μπορούσε να διευρύνει το, τη βάση δεδομένων του IMI, του Συστήματος Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς κάτι που θα διευκολύνει το διοικητικό διάλογο μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη η έκθεση γιατί πραγματικά παρέχει τροφή για σκέψη και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Well, Well, I, I we... Σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε και στο μέλλον και θέλουμε να σας συνδράουμε με πολιτική υποστήριξη. Αυτή είναι και η ιδέα της έκθεσης πρωτοβουλίας άλλωστε. Ε, κύριε Κορνέλης, ε, κύριε Δεγιόγκ, θέλετε να δευτερολογήσετε μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Ευχαριστώ. Θα έχουμε εκτενή συζήτηση και κατά την εξέταση των τροπολογιών. Κάποια καθησυχαστικά σχόλια. Όταν αναφέρθηκα στη μαύρη λίστα εννοούσα ότι στόχος μου στην έκθεση είναι να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ιδρύματα και τις κυβερνήσεις που ταλανίζονται από τέτοιες πρακτικές. Συμφωνώ ότι το να συντάξουμε μια μαύρη λίστα των επιχειρήσεων μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Γιατί ακόμη και αν καταδικαστούν οι μπορούν να αλλάξουν τον τίτλο τους ε, και να ξεφύγουν ούτως ή άλλως από το μαύρο κατάλογο, από τη μαύρη λίστα. Η αλλω απο το μαυρο όμως μαύρης ομως μαυρη λιστα με τις πρακτικές της αθέμητη, ε, αυτό είναι μια λύση που θα ήθελα να την εξερευνήσουμε και περαιτέρω. Γιατί τέτοιου είδου μέτρα και προτάσει θα είδαμε και στο Ολλανδικό Σημείο Επαφής Είχαμε μάλιστα πληροφορίες και κάποιες ε, εικόνες για το πώς ε, σας προσεγγίζουν τέτοιες ε, επιχειρήσεις. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έχουμε κάτι τέτοιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα συλλογικά έδικα μέσα, συλλογικές προσφυγές ή αγωγές, συναντήθηκα με τον κύριο Μίμιτς που είναι ο υποψήφιος επίτροπος για θέματα καταναλωτή και είπε ότι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σύσταση για τις συλλογικές αγωγές. Ε, αν θέλουμε κάτι, γιατί το θέμα της συλλογικών αγωγών το έχουμε αναφέρει σε πολλές εκθέσεις μας, ίσως θα πρέπει να το πούμε και με τις τροπολογίες. Πάντως, καλό θα ήταν είμαστε ρεαλιστικοί, θετικοί και σίγουρα οι τροπολογίες και των σχεδόν εισηγητών και των ε, ευρωβουλευτών θα βελτιώσουν την έκθεση. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε και θεσμικά όργανα και οργανισμούς, αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κατά των ε, θέμητων αυτών πρακτικών. Και φυσικά θα βρούμε πρόσφορο κοινό έδαφος και κοινέ λύσεις. Σας ευχαριστώ, λέει ο Ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή. 18 Ιουνίου η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα, το, θα τις εξετάσουμε αργότερα, ελπίζοντας να τις εγκρίνουμε στις 26, να εγκρίνουμε την έκθεση 26 Σεπτεμβρίου, μάλλον 25 Σεπτεμβρίου θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Οπότε 8-9 Ιουλίου θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για τις τροπολογίες, αν ε, έχουν ε, ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Και φαντάζομαι και η κυρία Μανφρέτ ε, θα μας ενημερώνει στο μέτρο που ανακύπτουν από τη μελέτη νέα στοιχεία και πληροφορίες. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσης διάταξης και θα περάσουμε σε μια γνωμοδότηση. που θα επιδώσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με θέμα τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικών δικαιωμάτων και χορήγηση αδειών πολλαπλή εδαφική ισχύω, ό,τι αφορά τα μουσικά έργα για επιγραμμικέ χρήσει στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω θερμά για την παρουσία του τη Μαρία Μάρτιν Πράτ, που είναι παλιά γνώριμο τη Επιτροπή Είναι αρμόδια, της, είναι τριματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Αγορά ε, για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Ο συντάκτη γνωμοδότησή μα είναι ο Τόιν Μάντερ. και οι σκιώδες ηγητές είναι η κυρία Βερχέν, ο κύριο Χόλτς από του σοσιαλιστές, δεν ξέρω αν η κυρία Στάιλερ θα μείνει. Πού πήγαν οι σκιώδες ηγητές ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Έχει καταρρεύσει το, το σύστημά τους. Εγώ θα εκπροσωπήσω την κυρία Μακλάρκιν και ο Κορνέλης Δε Γιόγκ ε, θα εκπροσωπήσει την ΚΟΕ. Σχεδόν έχουμε απαρτία των σχεδόν εισηγητών. Και μάλιστα με βαρέαν βαρών εισηγητές. Γύρω στις 200 τροπολογίε έχουν υποβληθεί για την γνωμοδότηση σου, Τόιν. Τι γνώμη έχει γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, πραγματικά αυτό ακριβώ δείχνει ότι για γνωμοδότηση ο φάκελο είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ισορροπία. Οι καταναλωτέ όμω, όπω γνωρίζουμε, εξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήματα σε αυτέ τι υπηρεσίε και η αδειοδότηση, η διαδικασία είναι αρκετά αργή, περίπλοκη και όχι διάφανη και αυτό που έχουμε ακούσει από την Επιτροπή στην ε, μελέτη αντικτύπου που έχει διεξάγει είναι ότι οι δικαιούχοι δεν παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, αυτοί που δημιουργούν τα έργα δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στην ουσία είναι πάρα πολύ καλή, είναι κάτι που το συζητήσαμε νομίζω τους τελευταίους μήνες ή πριν από δύο εβδομάδες τελευταία φορά. Εγώ κατέθεσα 50 διαφορετικές ε, τροπολογίες, τροποποιητικές. Αφού το συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα για την νομοθεσία σχετικά με τον ανταγωνισμό, όπου πρότεινα μία απόδειξη, μία ενιαία απόδειξη για να αποφύγουμε προβλήματα με νομοθετικά, νομοθετικής φύσης. Τη μία ενιαία απόδειξη την ε, άλλαξα, την τροποποίησα και τώρα έχω προτείνει απόδειξη από το κράτος ή την περιοχή τέλο πάντων στην οποία διαμένει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε γενικές γραμμές ε, με στήριξαν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι έχουμε περιθώριο για να συμβιβαστούμε και να μειώσουμε τον αριθμό των τροπολογιών, διότι πιστεύω ότι το σκεπτικό πίσω από τη βελτίωση της ε, εσωτερικής αγοράς για την διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων είναι κάτι τα πάρα πολύ σημαντικό. Τρία είναι τα σημεία τα οποία θέλω να συζητήσω. Είναι η διασυνοριακή συνεργασία καταρχάς. Εκεί έχω κάποιες τροπολογίες οι οποίες αφορούν μέτρα προστασίας Κρίμα που έφυγε και ο Ρομπέρ, γιατί τον αφορούν. Ε, και αναφέρονται επίσης και σε εξαίρεση του τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Επίσης η Σαμπίνε έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δει όμως ορισμένες τροπολογίες τι οποίες καλό είναι να διευκρινίσουμε. Για παράδειγμα, η 220. Εκεί γίνεται λόγος για ένα πουλ, για ένα συγκεντρωστικό σημείο. Αυτό τι θα είναι, θα είναι ε, κυβερνητικός οργανισμός, θα είναι υποχρεωτικό ή θα είναι ένας εθελοντικό οργανισμός στον οποίο θα συμμετέχουν ε, προαιρετικά. Θα μπορούσατε λοιπόν να μα το εξηγήσετε. Επίσης, Έχω δει κάτι που εγώ ονομάζω μέτρα προστασίας, προστατευτικά, δεν ξέρω αν είναι. Για παράδειγμα, η τροπολογία 107. Εάν δεν απλουστεύσουμε την αγορά και διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου. Τότε θα δημιουργήσουμε πάρα πάρα πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα στην νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε και πρέπει να το κοιτάξουμε πιστεύω. Επίσης, δεν είμαι υπέρ της ε, εξαίρεσης τομέων όπως ε, οπτικοακουστικός. Πιστεύω πως ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με πνευματικά δικαιώματα, τα οποία πολλές φορές ε, και όλο και περισσότερο στις μέρες μας γίνονται στο διαδίκτυο και δημοσιεύονται εκεί. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν θέλω λοιπόν να εξαιρέσω τομείς και να τους αποκλείσω από την πρόταση. Αυτά εν ολίγης για τώρα. Την επόμενη εβδομάδα σκοπεύω ή την Τετάρτη ή κάποια άλλη μέρα να συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε εάν μπορούμε να συμβιβαστούμε και μετά από τη σημερινή συζήτηση στην οποία ε, θα ήθελα κιόλας να καλέσω και τους υπόλοιπους ε, που κατέθεσαν τροπολογίες να το συζητήσουμε και να μου τις απόφα να, τις, αποφασίσουμε πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση την επόμενη εβδομάδα και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μετά και μετά να στείλουμε τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έτσι ώστε να συμπεριλάβουν στη δική τους έκθεση τις ε, πτυχές της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως τον Τόιν Μάντερς, ο οποίος ε, έφυξε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, ιδιαίτερα την δίκαιη αμοιβή, την ε, διαφάνεια, του ε, δικαιούχου και που προσπάθησε να πλουστεύσει την διαδικασία αδειοδότησης, ε, κάνοντάς την αποκεντρική σε πολλαπλές περιφέρειες. Ήδη το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για το one-stop shop, για την διαδικασία της της ενίας, ενίας θηρίδας. Είναι λίγο δύσκολο να, το, να πραγματοποιήσουμε αυτή τη λύση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πάρα πολλές επιπλοκές. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι διαφάνεια. Διαφάνεια για τους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή μια άδεια για τις τράπεζες δεδομένων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως κατά την άποψή μου να είναι ή ή ακόμα και παγκόσμιες Επίσης θα χρειαστεί για αυτές τις τράπεζες δεδομένων να συσταθεί ενδεχομένως ένας ε, παγκόσμιος ε, κεντρικός οργανισμός διαχείρισης αυτών των τραπεζών δεδομένων ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα, ποια δικαιώματα ε, αφορούν, ποια είναι η δομή στην τιμολόγηση των αδειών. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να συζητηθούν. Υπάρχουν επίση ένα-δύο σημεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε γιατί μπορούν να είναι ενδεχομένω προβληματικά. Καταρχά, η ε, πρόταση για διαγραφή ε, του οτιδήποτε αναφέρεται στην. Ε, οδηγία παροχή υπηρεσιών. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πολύ ισχυρή και αυστηρή νομοθεσία που διέπει αυτόν τον τομέα. Κάποια άλλα κράτη καθόλου. Υπάρχει λοιπόν νομοθεσία που εμποδίζει την εστρέβλωση της αγοράς σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και έχουμε πάρα πολλέ διαφορέ, αλλά πιστεύω πω σίγουρα μετά από συζήτηση θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα, διότι ο καθένα μα θα συνεισφέρει με την δική του διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αδειοδότηση, τη χορήγηση άδειων για, τα, για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των ε, κατόχων των δικαιωμάτων αυτών ανά κράτος μέλος και να προσπαθήσουμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλες αυτές ε, τις διαφορετικές νομοθεσίες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο. Τώρα, όπως είπατε, αυτά τα pools, αυτές οι συγκεντρώσεις διαδικτυακών δικαιωμάτων, να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν προαιρετικά διαφορετικά πιο τοπικοί οργανισμοί και αυτό ίσως θα διευκολύνει το έργο της ε, διαδικασίας αδειοδότησης. Χρειάζονται φυσικά ε, να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τους, πρέπει να οργανωθούν, να έχουν κάποια, κάποια δομή, κάποια διοικητικά όργανα. Αυτό είναι όντως κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, διότι η διασυνοριακή συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ περίπλοκο. Ιδιαίτερα όταν κάποιο θέλει να αποκτήσει ε, μία άδεια πολυπεριφερειακή που να ισχύει σε παραπάνω από ένα κράτος μέλος. Αυτές, ε, αυτή η λύση λοιπόν του, του πουλ είναι περίπλοκη, αν και θα ήταν καλή αν ήταν εφικτή. Επίση, κάτι που θεωρώ καλό και πολύ χρήσιμο είναι οι προδιαγραφές για την διαφάνεια για τις εταιρείε ε, αξιολόγησης και διαχείρισης των δικαιωμάτων και πιστεύω πως πρέπει να έχουν την δυνατότητα οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, αλλά και όχι μόνο και οι νομικοί που τους εκπροσωπούν να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησης, συλλογικής εκπροσώπησης. Διότι σίγουρα ένας καλλιτέχνης μόνος του ή ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να έχει τόσο καλή εκπροσώπηση όπως μια οργάνωση, μια ένωση. Και φυσικά όταν ε, σε μια περίπτωση διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων κάποιο έχει να κάνει με μια οργάνωση παρά με έναν ε, μόνο ιδιώτη, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σε γενικέ γραμμέ ε, πιστεύω πω θα βρούμε καλού ε, συμβιβασμού και θα έχουμε έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ. Όπως Είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, όλοι θέλουμε διαφάνεια, όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι καλλιτέχνες, οι δικαιούχοι παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν και πιστεύω θα βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες που είναι προβληματικές και όλες είναι δικές μου, δυστυχώς. Ε, it's number 94 213 και 242. Η ίδια ιδέα από πίσω είναι πάντα. Η πρόταση της Κομισιόν λέει οι εταιρείε που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος. Εγώ ε, το έκανα που δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος μέλος. Η ιδέα μου ποια ήταν. Να μην μπορούν να καταχωρούνται αυτές οι εταιρείε σε διάφορες χώρες αυτές εταιρείε συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων. Αλλά το... Γιατί δεν θέλουμε και το κάθε κρατός να, πρίνει, να πρέπει να δίνει άδεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Δυστυχώς... Νομίζω ότι με τη διατύπωσή μου δεν διευκολύνω τα πράγματα. Τη αποσύρω και ζητώ συγγνώμη για την κακή Κάτι γενικότερο. Αυτή η ιδέα της ενιαίας θηρίδας. Ο κύριος Μάντες το πρωτοανέφερε. Καλή ιδέα. Έχετε και οι δύο δίκιο. Α, θέτει θέματα ανταγωνισμού και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Η κυρία Φερχόη είπε εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση. Αν εγώ ήμουν μέλος μιας τέτοιας ε, εταιρείας λογικής διαχείρισης, θα προτιμούσα ένας δικηγόρος, ένας επαΐοντας να με εκπροσωπήσει και όχι ένας καλός κιθαρίστας, ας πούμε, που είναι άσχετος από νομική. Έχω υποβάλει μία τροπολογία ε, σχετικά και πιστεύω ότι θα βρούμε καλούς συμβασμούς και για αυτό το σημείο. Αποκλεισμό των οπτικοακουστικών. Όχι. Υπάρχουν ε, προβλήματα σε αυτό το τομέα, έλλειψη διαφάνειας κτλ. Αλλά ο οπτικοακουστικός οποιος, οποιοδήποτε άλλο τομέα είτε έχει αυτά τα προβλήματα και τότε θα πρέπει να, τα, να εντάξουμε αυτές τις τρο... να τον εντάξουμε μάλλον αυτόν τον τομέα, είτε δεν έχει αυτά τα προβλήματα, οπότε... Και τότε δεν έχει σε άλλο τομέα, οπότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Για μένα, Η πιο σημαντική τροπολογία είναι αυτή που υπέβαλε για το άρθρο 12.2. Αν η εταιρεία δεν μπορεί να βρει τον κατάλογο με τους δικαιούχους, δεν πρέπει να κρατάει τα λεφτά. Γιατί ε, έτσι όπως έχουμε τη διατύπωση τώρα, είναι σαν τους δίνουμε τη δυνατότητα να μην ψάχνουν για αυτούς. Εντάξει, καλέ είναι οι δικέ τους ε, πολιτιστικές δραστηριότητε, αλλά ε, τους δίνουμε κίνητρο να μην ψάξουν να τους βρουν αυτούς του δικαιούχου. Τα λεφτά πρέπει να πάνε ε, στους δικαιούχους αυτούς που γράψανε αυτά τα έργα, όχι σε κάποιους άλλους που ανήκουν σε αυτές τις εταιρείες σε αυτές τις εταιρείες ε, διαχείρισης λογικών δικαιωμάτων. Στην οδηγία για τα ορφανά έργα αποφασίσαμε ότι οι βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Europeana που ψηφοποιούν τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το βάζουν online. Και εκεί κάποια στιγμή εμφανίζεται ο εγγόνο κάποιου δικαιούχου, α πούμε. Εντάξει, να πάρει την αποζημίωση. Αλλά αυτά τα λεφτά που έχουν ε, συλλεχθεί θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, για αυτή την ψηφιοποίηση κτλ. Γιατί θέλουμε όλοι αυτή η πολυπίκυλη ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να είναι διαθέσιμη σε όλους αλλά μπορεί ο διάβολος να κρύβεται τις λεπτομέρειες και με αυτές τις διατάξεις να το παρεμποδίζουμε. Να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά δηλαδή ε, για να ε, θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις, τις απαιτήσει που βαραίνουν τις βιβλιοθήκες να πληρώνουν τέτοια δικαιώματα. Αυτά, κύριε Άνστρομ. Θα αντικαταστήσω τώρα τη σκιώδη μας την κυρία Μακλάρκιν, που είναι και σκιώδης και στην Ομπική Επιτροπή. Έχει πολλές γνώσεις για το θέμα αυτό. Όπως λοιπόν και οι υπόλοιποι σκιώδης ηγητές και η κυρία Μακλάρκιν ευχαριστεί τον Τουαν Μάντερς θερμότατα για τη γνωμοδότησή του και ήταν πολύ επιλεκτική στην κατάσταση των τροπολογιών γιατί συμφωνεί με τη βασική δομή της γνωμοδότησης και δεν ήθελε να την διαταράξει. Τι προβληματίζεται η κυρία Μακλάρκινγκ και ελπίζω, ελπίζει στην συμφωνία με του εισηγητού. Δεν συμφωνεί με το γεγονός ότι ο εισηγητή θέλει να διαγράψει την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει τα κράτη-μέλη να αποκλεί τις μικρές εταιρείες ε, συλλογών από υπερβολικό άχθος. Είναι λογική αυτή η πρόταση να απολαγούν οι μικρές επιχειρήσεις από τέτοιο άχθος. Γιατί λοιπόν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ε, που μπορεί να είναι και ειδικευμένες στον τομέα τους να ξεφεύγουν από αυτή τη γενική διάταξη δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη της κυρία Μακλάρκιν. Επίσης ε, θα υποβάλει τροπολογίες για να ισχύσει αυτό το σύστημα χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύω. γιατί σε αυτό το τομέα ακριβώς ε, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ε, ιστοσελίδες πολλαπλής ε, εδαφικής ισχύω ε, και σε πολλές περιοχές. Έχει νόημα λοιπόν. Επίσης, το θέμα της συλλογής κονδυλίων για κονδύλια που δεν έχουν διανεμηθεί ή ε, προσημειωθεί. Νομίζω η κυρία Μακλάρκη θα μπορούσε να γίνει απελευθέρωση αυτών των κονδυλίων για ορθολογική τους χρήση. Η κυρία Μακλάρκινγκ ε, ζητά με τις τροπολογίες της ε, συνεργασία μεταξύ των των επιχειρήσεων συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων ε, και πιο, απλών, ε, πιο απλής αποστολής λογαριασμών για τους πολίτες, για τους πελάτες. Θα στείλω στον κύριο Μάντερς ε, τη σημειώση μου για να έχει και γραπτό στη σοφία της κυρίας Μακλάρκινς. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντε και βλέπω ότι έχει φτάσει και η σκιώδη ηγέτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, που δεν έχει βάλει ακόμη τα ακουστικά τη ακούσει αλλά ούτε άκουσε τη ζήτηση μέχρι τώρα, γιατί έγινε μια ε, τροποποίηση τη σειρά των διαφορών σημείων, αλλά είναι σημαντικό που ήρθε ο σκιώδη ηγετής από, το, από τους σοσιαλιστές. Βέβαια, δεν είναι την τελευταία στιγμή που αλλάξαμε το χρονοδιάγραμμα. Πριν από δύο μέρες λάβατε την αλλαγή του σημείο της ημερήσιας διάταξη. Ε, θα δώσω πρώτο λόγο στον κύριο Ντεγιόνκο, ώστε να έχετε το λόγο να καθίσετε ήρεμα και να μπορέσετε να σχολιάσετε τα Κύριε Πρόεδρε, το... και εγώ και η βοηθή μου στρωθήκαμε και συγκεντρώσαμε, καταρτήσαμε δεκάδες τροπολογίες, γιατί μιλήσαμε και με πολλούς ενδιαφερόμενους, αλλά στο μεταξύ έλαβα το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Μάντερς και ε, ξεπλάγει πολύ θετικά, γιατί ε, το ενιαίο τιμολόγιο είναι η λύση με την οποία συμφωνούν ε, σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό σημείο φετηρίας αυτό για μας. Και ελπίζω να διαφυλαχθεί αυτή η αρχή του ενιαίου τιμολογίου, γιατί πραγματικά ανταποκρίνεται σε αιτήματα μεγάλου φάσματος εμπειρογνωμόνων. Τώρα, οι τροπολογίες μου τελικά λοιπόν ε, θα είναι πολύ λιγότερες από αυτές που είχα σχεδιάσει ε, στην αρχή. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και προσβλέπω σε στενή συνεργασία και με τους υπόλοιπους καθηγητές και με τον εισηγητή μας γι' αυτό. Θα καταθέσω τροπολογίες ε, για το πεδίο εφαρμογή φυσικά. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τον ορισμό ώστε να περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις και τις εμπορικές φυσικά. Γιατί αυτό που δεν μου άρεσε και πολύ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η ιδέα ότι οι, εντάξει, εμπορικές οργανώσεις και οι εμπορικοί φορείς και το πρόβλημα έχουν οι ενώσεις μη εμπορικό χαρακτήρα. Το πρόβλημα με τις ενώσεις υπάρχει και νομίζω ότι είναι πολύ η υπερβολική γενίκευση να λέμε ότι αν κάποιο ε, ε, αποκαλεί την επιχείρησή του τον εργάζεται στην εμπορική δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει και εδώ να δούμε τι προποθέσει που θα εφαρμόσουμε. Στο πρότυμα της Το πρότυμα τη Ευρωπαϊκής... Ε, πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ισχύει και για του υπόλοιπου φορεί, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Δεύτερον, κάτι που ισχύει και για τη μουσική και για άλλου τομεί. Εκεί που έχουμε συγκεκριμένου θύλακε, κλειστέ αγορέ, νη, ε, για, για, διά, για περιεχόμενο, για συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Και νομίζω η πρόκληση για μας είναι να εκπροσωπήσουμε όχι το βασικό, το συνηθισμένο ρεπερτόριο, αλλά και ρεπερτόριο ειδικό, συγκεκριμένων θυλάκων, νης. Επίσης, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε και σε συγκεκριμένες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες η ομάδα μου θεωρεί ότι θα πρέπει αυτή η επιλογή να παραμένει ανοιχτή ε, για τις οργανώσεις, γιατί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν πάντα σαφές για το σημείο αυτό. Μερικές φορές αναφέρεται, η δυνατότητα μερικές φορές παραλείπεται, αλλά για μας είναι προτεραιότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Φερχέιεν για το δίκαιο του ανταγωνισμού, γιατί αφενός θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα αδειοδότησης πολλαπλής εδαφικής ισχύω για να δημιουργήσουμε ένα είδος αγοράς, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να προωθήσουμε και τον ανταγωνισμό, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων. θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή. Και εδώ περισσότερο θα πρέπει να συνεργαστούμε παρά να αφήσουμε το δίκαιο ανταγωνισμού να στρεβλώσει τη συνεργασία ή να την καταστήσει αδύνατη. Νομίζω αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και είναι πολύ καλό σημείο αφετηρία η έκθεση του κύριου Μάντερς για τα θέματα αυτά. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στι συμβαστικέ λύσει, γιατί ήδη η αφετηρία, παραλαμβάνω, ήταν πολύ καλή. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ. Έχω επίσης την ίδια θετική εκτίμηση. Χαιρετίζω την πρόταση για την οδηγία αυτή, η οποία αντικατοπτρίζει πραγματικά τις εξελίξεις στον ψηφιακό χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ισχύουσα κατάσταση για τους καλλιτέχνες δίνει πάρα πολύ μεγάλη νομική ασάφεια. Κανείς δεν ξέρει πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει μία έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικά οργανωμένης ε, διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχύον σύστημα εκτός από όλα αυτά είναι και πολύ περίπλοκο. Και το περίπλοκο αυτού του συστήματος πραγματικά εμποδίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη στον χώρο αυτό. και είναι προς το συμφέρον όλων μας να εργαστούμε για την απλούστευσή του. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες, έχω υποβάλει και εγώ κάποιοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε ε, πολλαπλή ε, ισχύω. Πιστεύω πως αυτό θα προσδώσει διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία, θα πλουστεύσει την ε, διαδικασία. Και είναι σημαντικό να υπάρχει λοιπόν αυτή η χορήγηση αδειών σε πολλαπλά επίπεδα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ένα κράτος μέλο αρνείται τη χορήγηση άδεια και αυτό εμποδίζει την πνευματική δημιουργία και την εξάπλωση ενός προϊόντος σε ακόμα περισσότερα περισσότερα τώρα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιορίσουμε το εύρος Επίσης, το θέμα της αμοιβή πρέπει να ρυθμίζεται με καλύτερο τρόπο. Οι προθεσμίες θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι συντομότερες οι προτάσεις της κυρίας Φερχόν με βρίσκουν σύμφωνο διότι οδηγούν σε μια εκδημοκρατήση της διαδικασίας και πραγματικά αυτό θα βοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για την καλή δουλειά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσε και συμμετείχαμε ενεργά στην ε, έκθεση αυτή. Ελπίζω οι προτάσεις μας να συμπεριληφθούν και οι προτάσεις οι δικές μου ιδιαίτερα όσον αφορά τις αμοιβέ και το ζήτημα του ποιος αποφασίζει για τις αμοιβέ και πώς αυτές γιατί και για το ύψος του και πώς αυτές κατανέμονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος εκτός από τους κύριους εισηγητές να συμμετέχει στη συζήτηση. Όχι. Τότε θα καλέσω την Μαρία Μάρτιν Πράτ να μας εκθέσει τις δικές της απόψεις για τις τροπολογίες από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που έχω αυτή την ευκαιρία. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντερς για τη δουλειά που έχει κάνει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μέλη, και κοιόδης συζητητέ, για το σύνολο των 242 τροπολογιών στην έκθεση αυτή, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αρχίσω λέγοντας ότι στηρίζω απόλυτα ορισμένες από τις αρχές που ανέφερε ο κύριος Μάντερς και οι σκιώδες εισηγητές ε, στις παρεμβάσεις τους ε, συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι η σημασία της βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, την οποία καλύπτει η οδηγία, η σημασία της βελτίωσης της διαφάνειας, η συμμετοχή και ο, ε, η δυνατότητα ελέγχου των εκατόχων των δικαιωμάτων και η σημασία της απλούστευσης διαδικασίας διοδότησης και απλούστευσης της ζωής των κατόχων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να γίνονται σεβόμενα το δίκαιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από την Επιτροπή αυτή εδώ από το να βοηθά στην βελτίωση των συνθήκων για τους καταναλωτές. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα τα οποία είναι προβληματικά. Στα ψηλά γράμματα κρύβονται τα σημαντικά όπως ξέρετε. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία πιστεύω πως θα πρέπει να έχετε σοβαρά υπόψη τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με εμά να τα έχετε υπόψη σας καθώς συντάσσετε την έκθεσή σας και καθώς ενσωματώνετε τις τροπολογίες στο κείμενο. Καταρχάς, η πρώτη μας ανησυχία αφορά 13 τροπολογίες τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει μη φιλικές προς την εσωτερική αγορά, μάλλον αχθρικές θα έλεγα. Κύριο Έμστρομ, δείχνοντας αλληλέγγυο πνεύμα, μας είπε ότι αποσύρει τρεις από τις δικές του τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ευχαριστεί για αυτό, διότι πραγματικά είχε θίξει ορισμένα προβληματικά σημεία. Τη αναφορά στην ανάγκη ε, ελεγχόμενων δραστηριοτήτων σε κράτη-μέλη τα οποία έχουν ήδη θεσπίσει δική τους νομοθεσία και η ενεργή ή ανενεργή διάσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιους ότι δεν είναι τόσο φιλική προς την ενιαία αγορά, αλλά θέλει να προσδώσει τον έλεγχο κυρίως στα επιμερούς σε κράτη-μέλη. Και όταν μιλάμε για τη χορήγηση αδειών σε πολλές σε αυτό θα δυσχεράνει την ε, χορήγησή τους. Παρακαλώ, εκτός μικροφώνου. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά ελπίζω και ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές να έχουν υπόψη τους ε, τη χώρα προέλευσης των ε, δικαιωμάτων αυτών. Το έχουμε ήδη συζητήσει με την κυρία Φερχάικεν. Αλλά με όλο το σεβασμό να πω ότι ορισμένες τροπολογίες όπως οι 107 περιέχουν κάποια στοιχεία όπως για παράδειγμα η αναφορά σε, μια, σε ένα σημαντικό μερίδιο του ρεπερτορίου ενό καλλιτέχνη σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, τότε το κράτος μέλος αυτό θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των πνευματικών του δικαιωμάτων, ακόμα και αν αυτός ο καλλιτέχνης έχει εγκατάσταση νόμιμη σε κάποιο άλλο. Καταρχάς αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο ποσοστό ενός ρεπερτορίου θεωρείται σημαντικό. Τι θεωρείται σημαντικό και έπειτα. Ας υποθέσουμε ότι μια γαλλική εταιρεία χορηγεί σε ένα χρήστη, είτε αυτός είναι μεγάλος, είτε είναι το Spotify, είτε είναι κάποιο site για να κατεβάζεις υλικό, είτε κάποιος μικρός. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή η γαλλική, ο γαλλικός οργανισμός χορηγεί σε αυτόν τον χρήστη μια, χορηγή, μια άδεια πολλαπλής εδαφικής ισχύω. Τότε τι θα γίνει εάν η άδεια αυτή αφορά υλικό το οποίο διατίθεται κυρίως στη Γερμανία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Τι θα γίνει, αυτό το σημαντικό μερίδιο λοιπόν του υλικού, του καλλιτεχνικού υλικού θα διέπεται από γαλλικούς νόμους, από γερμανικούς νόμους, ποιος θα ελέγχει, η Γαλλία ή η Γερμανία. Πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό κιόλα είπα ότι αυτή η τροπολογία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μη φιλική προς την εσωτερική αγορά και θα ενδεχομένως καταστρέψει αυτό που προσπαθούμε εμείς να χτίσουμε. Τώρα, όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού. Μια χαρά είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού. Είναι καλό για τους καταναλωτές, είναι καλό για την ανάπτυξη της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει έρθει εδώ με όπλα στη φαρέτρα τη με ένα σωρό νομοθετήματα για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συλλογικές ε, εταιρείε που να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος, ε, να αντιπροσωπεύουν πολλού καλλιτέχνε και να μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα του χρήστες. Δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια επιταγή και να δώσουμε το και χωρίς να ρωτήσουμε καν γιατί. Δυστυχώς όχι, δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τα άρθρα 101 και 102 της συνθήκης. Είναι αδύνατον. Δεν θα ήταν καλό. Και εδώ συμφωνώ και με την κυρία Φερχόγγεν, ε, όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε. Φυσικά μπορούμε να συνεργαστούμε. Καταρχά οι αμοιβέ ε, συμφωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Κανείς δεν απαγορεύει να υπάρχουν ε, συμφωνίες τέτοιου είδου. Εάν προσπαθείτε να συγκεντρώσετε τις πρακτικές με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι άλλο από το να λέτε ότι θέλουμε να συγκεντρώσουμε τι τιμέ στα εκάστοτε κράτη-μέλη και να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο κατάλογο αναφορά. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Επίση, αναφέρατε αυτή την παγκόσμια τράπεζα δεδομένων όσον αφορά το ρεπερτόριο και αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά στι τροπολογίε δεν μπορούν να περιέχουν κάτι τέτοιο το οποίο θα έρχεται σε άμεση σύνδεση με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τώρα, όσον αφορά τα Του τους ε, αναμεταδότες, τα κανάλια, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Στο άρθρο 33 της δικής μας πρότασης αναφερόμαστε ειδικά σε αυτούς τους οργανισμούς και όλες τις βοηθητικές και συνοδευτικές ε, δραστηριότητες που σχετίζονται λοιπόν με, τις, ε, με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, με τα κανάλια και όλους αυτούς ε, τους οργανισμούς μετάδοσης. Αυτό πιστεύουμε, αυτοί θα υποφεληθούν από αυτήν την άδεια πολλαπλής εδαφικής ισχύω, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη το άρθρο 33 Εάν μια άδεια που έχει χορηγηθεί σε κάποιον οργανισμό μετάδοσης, γιατί να πρέπει να περιπλέξουμε τα πράγματα δημιουργώντας ε, αυτό το συλλογικό, αυτή τη συλλογική μορφή αδειών. Μετά υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες που συνδέονται με το άρθρο 5 ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο. Οι οποίες τροπολογίες μου φαίνεται πως θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία των κατόχων δικαιωμάτων. Να και να επαναλάβω, δεν θέλουμε μια οδηγία που να δίνει λιγότερη ελευθερία στους κατόχους των δικαιωμάτων. Θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερη ελαστικότητα, περισσότερες επιλογές. Έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανάγκες για ισορροπία και τις ανάγκες για μια συλλογική κοινότητα, για παράδειγμα τις 114 και 115, αυτές τις τροπολογίες είναι προβληματικές, διότι έτσι αφαιρούν τα δικαιώματα επιλογών από τους κατόχους των δικαιωμάτων αυτών. Πρόεδρε, τώρα κάτι τελευταίο σχετικά με τους εμπορικούς ε, φορείς. Πρέπει να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε για αυτούς. Τι εννοούμε. Υπάρχουν πολλά είδη εμπορικών φορέων. Για παράδειγμα, οι ατζέντιδε, ας πούμε, των καλλιτεχνών και αυτοί θεωρούνται εμπορικοί φορείς. Είναι εταιρείε οι οποίες βοηθούν τους καλλιτέχνες ή τους δημιουργούς να λάβουν τα χρήματα τα οποία ε, αναλογούν στην εργασία τους. Κύριε Μάντες, τα ξέρετε από τη δική σας χώρα. Και αυτοί κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, διότι, όπως είπατε κι εσείς, ο καλλιτέχνης είναι καλός κιθαρίστας, αλλά εκείνοι είναι καλοί διαχειριστές και τον βοηθούν να λάβει τα χρήματα που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν το να βάζουμε αυτούς τους φορείς στο, ίδιο καλάθι με το κράτος και με άλλες υπηρεσίες πιστεύουμε και μάλιστα χωρί να ζητούμε συγκεκριμένη εντολή, χωρί να ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητε, χωρί να έχουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι στην διαδικασία. Πιστεύουμε πω αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξανασκεφτείτε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι άλλο το να δημιουργήσουμε, το να θέλουμε μάλλον να δημιουργήσουμε ίσους όρου, και είναι άλλο να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε έναν κανονισμό με τον οποίο θα μείνουν έξω αυτοί οι σημαντικοί παράγοντες. Αυτές λοιπόν είναι ορισμένες από τις ανησυχίες μας. Να επαναλάβω ξανά, ξα, ξανά τις ευχαριστίες μου για την εξαιρετική δουλειά του συγητή και, αυτή, και αυτής της Επιτροπής και να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει ό,τι εσείς χρειάζεται. χρειάζεστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την πολύ εξαντλητική απάντηση. Κύριε Μάντες, έχετε να προσθέσετε κάτι. Μετά το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε και χρόνο. Γρήγορα παρακαλώ. Τρώτε από την επόμενη έκθεσή σας το χρόνο. Σύντομος θα είμαι. Η ενιαία θηρίδα, όπως είπε η συνάδελφος, είναι μια εθελοντική συνεργασία, εξασφάρει μια εθελοντική συνεργασία χωρίς ε, κυβερνητικό έλεγχο. Η κυβέρνηση ελέγχει την ομοθεσία, όχι τη συνεργασία των εταιριών. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν έτσι τη λύση. Ο Κρίστιαν έκανε μια πολύ αστεία παρουσίαση. Ευχαριστώ που μας απέστησες και τις τροπολογίες σου. Μάλκομ. Να σου διευκρινίσω γιατί διέγραψα τις μικρότερες εταιρείες συλλογής δικαιωμάτων. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Αν εξαιρέσει τις μικρές, τότε μπορεί οι μεγάλες να διρεθούν σε πολλές μικρές και να παρακάμπτουν την νομοθεσία. Εγώ είμαι δικηγόρος, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το σημείο αυτό. Γι' αυτό το διέγραψα. Εν συνεχεία το να δημιουργήσουμε ένα ταμείο. Είμαι κατά, γιατί είναι ακίνητρο. για να κρατάνε τα λεφτά. Ποιο έλεγχε τα λεφτά, ποιο κρατάει τα λεφτά, πώ θα ξοδευτούν. Χρειαζόμαστε και άλλε οργανώσει. Γι' αυτό είπα να διαγραφεί το ταμείο. Δεν θέλω να δημιουργηθεί το ταμείο και να μένουν και τα λεφτά. Ίσως ε, θα πρέπει να βρούμε και έναν σκοπό για τον οποίο ξοδεύονται αυτά τα λεφτά. Το δημοκρατικό, η δημοκρατικότητα των εταιριών. Ναι, να το βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι είναι θελοντικά συστήματα αυτά. Εσύ ως καλλιτέχνης μπορεί να ενταχθείς. Εάν δεν σε αρέσει αυτή η εταιρεία, επιλέγεις μια άλλη. Νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται με αυτή την πρόταση. Ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός έχει μια επιλογή. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εταιρεία που προτιμά να τον εκπροσωπεί και να συλλέγει τα δικαιώματά του. Είναι δυνατό λοιπόν με αυτή την πρόταση. Και οι εταιρείε δεν θα πρέπει να ελέγχουν του καλλιτέχνε, του δημιουργού, θα πρέπει να του διευκολύνουν βασικά. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να συμβιβαστούμε. Uh, Θέλω να καλέσω τους κοιόδες εισηγητές την ε, Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, να συνεδριάσουμε μία-μία μισή ώρα για να δούμε πώς μπορούμε να συμβιβαστούμε. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, δηλαδή. Αν σας αρέσει αυτή η πρόταση, θα σας στείλω και μία πρόσκληση. Πότε και πώς ακριβώς θα συναντηθούμε. Θέλω να συναντηθούμε, θέλω να συνεργαστούμε για να υποβάλω μια καλή πρόταση που θα την υποστηρίξουν όλοι, ακόμα και οι Κομισιόν. Θα την ανεχτεί έστω. Ευχαριστώ. Αν τα πάτε καλά, στις 17 Ιουνίου θα έχουμε ευκαιρία να δούμε τις συμβαστικές τροπολογίες και στις 18 θα ψηφίσουμε. Γιατί το όριο είναι η 9η Ιουλίου με την ενεργητικότητά σας και το ζήλο σας είμαι σίγουρος και με έτσι τη χαλαρότητα που σας διακατέχει θα φτιάξετε πολύ κομψούς ε, συμβασμούς χωρίς δυσκολίες. Α, σας ευχαριστώ για τα κοπλιμέντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. Πάμε τώρα στη δεύτερη έκθεση Μάντερς. Πολλά, δουλειά σας βάζουμε. Είναι μια νομοθετική έκθεση. Είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Κύριε Μάντες, με ακούτε? Παρακαλώ, προσέξτε με. Τη δουλειά με τους σκιώδεις συζητητές θα την αρχίσετε αργότερο, όχι τώρα. Βρήκαμε και πότε θα συναντηθούμε, λέει ο κύριος Μάντες. Δεν σας είπα να πάρει το λόγο ακόμα. Ο κύριος Γκούχα, ελπίζω να είπα καλά το όνομά του, τον, τον ε, ε, καλωσορίζω από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκτα. Προϊόντα, αγορά και εφαρμογή. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μονάδα σας. Α, είναι Γενική διαθέση Επιχειρήσεων. Εγώ νόμιζα ότι είναι Γενική διάθεση Μάρκετ, έτσι μου γράφεται. Για την απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτο εντό ενία αγοράς. Θα θυμάστε ότι αυτό ήταν από τις μεγαλύτερε ανησυχίε των πολιτών για την ενία αγορά. Ζήτησαμε από τον Μισελ Μπαρνιέ ένα έγγραφο και αυτό εντοπίστηκε ως η μείζωνα ανησυχία. Η Κομισιόν λοιπόν ε, κράτησε το λόγο της να δώσει συνέχεια και τώρα εμείς νομοδοτούμε επ' αυτού του κειμένου και θέλουμε βεβαίως αυτές τις ιδέες να τις κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα κράτη-μέλη και να υιοθετήσουν αυτό το κείμενο και να το σεβαστούν. Θα ακούσουμε λοιπόν την έκθεση Μάντερς. Προτείνετε να το κάνουμε αυτό. Αν θέλετε, παρουσιάστε μας την έκθεσή σας. Ο κύριος Καράς είναι σκιώδης κυρία Στάιλ είναι εδώ, κυρία Ριούλε είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ πάντα. Από ό,τι φαίνεται η ομάδα των σκιωδών ε, εισηγητών είναι ντούρα. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω να... Έγραψα την έκθεσή μου. και έχει κάποια σημαντικά σημεία. Κατά να άποψή μου είναι σημαντικό τα οχήματα να ταξινομούνται εκεί που χρησιμοποιούνται. Είναι βασικό αυτό. Γιατί έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τον έλεγχο. Για διάφορους λόγους λοιπόν και λόγω διαφοράς στη φορολογία είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι γίνεται με τα κινητά παρακαλώ. Έχουμε ορφανό τηλέφωνο με στην αίθουσα. Ακούγεται και στο διαδίκτυο ο ήχος του. Μάλλον κάποιος έβαλε το, το ξυπνητήρι του για να ξυπνήσει όταν εσείς μιλήσετε. Είναι δύσκολος ο τελικός στόχος να υλοποιηθεί πάρα αυτά, αλλά με τις μοντέρνες ε, τεχνικές μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επαναταξινόμηση όχι σε υπόθεμα χάρτου, αλλά ηλεκτρονικά. Αυτό τι σημαίνει βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε όλες τις εθνικές βάσεις δεδομένων, αλλά θα τις συνδέσουμε με το Ιουκάρις. Υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων, θα τις συνδέσουμε λοιπόν μέσω του Ιουκάρις και θα έχουμε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που θα είναι το άθροισμα των εθνικών βάσεων δεδομένων. Τέλειο αυτό θα ήταν. Και έτσι θα είναι σαφές πότε αρνούμαστε την είσοδο ενό οχήματος σε ένα κράτο μέλο. Ε, ε, Υπάρχουν εταιρείε μεταφορών που μου έκαναν το εξή ε, ερώτημα. Έχουν καταστήματα ή θηγατρικέ σε διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουν κοινή αντιμετώπιση. Για αυτές τις εταιρείε προτείνω να μην έχουμε τους εθνικούς κωδικούς, γιατί εδώ υπησέρχεται η εθνική νομοθεσία. Δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Θέλουμε να δώσουμε δυνητικά την, τη δυνατότητα κάποιος να επιλέξει τα εθνικά του χρώματα. Εμείς έχουμε άσπρο μαύρο στην Ολλανδία, στο Βέλγιο άσπρο κόκκινο, μαύρο και κόκκινο στη Γερμανία, θέλω ο καθής να μπορεί να επιλέγει είτε την, ε, τα εθνικά χρώματα είτε τα ευρωπαϊκά. Αυτό είναι βολικό για τις ε, εταιρείε μεταφορών. Αν θέλουν να μην χρησιμοποιούν τα εθνικά χρώματα. Αλλά εγώ και, εγώ ίδιος προσωπικά θέλω να δείχνω ότι είμαι και Ολλανδός αλλά και Ευρωπαίος με τα χρώματα. Τα, τα πιστοποιητικά επίσης προσωρινής ε, ταξινόμησης. Υπάρχει η γερμανική οργάνωση ιδιοκτητών αυτοκινήτων που λέει ότι έχει πολλά προβλήματα εδώ. Θέλουμε κοινέ προσωρινές πινακίδες και σε όλη την Ευρώπη τα χρώματα να είναι τα ίδια, ούτω ώστε οι αστυνομίε σε όλα τα κράτη-μέλη και οι αρχέ γενικά να βλέπουν αμέσω ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει προσωρινέ πινακίδε, όχι μόνιμε, και να το αναγνωρίζουν. Κάτι άλλο που έκυψε στην ακρόαση είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα κατά τη απάτη. Πώ? Χρησιμοποιώντα τι έξυπνε κάμερε γίνεται και εισάγοντα επίσης τσιπάκια και στις πινακίδες και στο ίδιο το αυτοκίνητο. Ναι, να... Αν αγοράζει δηλαδή μία πινακίδα, θα έχει ένα τσιπάκι RIVD και παράλληλα θα έχεις και ένα αυτοκόλλητο που επίσης εμπλέκει ένα, έχει ένα τσιπάκι. Επομένως, η πινακίδα και το αυτοκίνητο μέσα από αυτό το τσιπάκι συνδέονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε άσχετο αυτοκόλλητο ας πούμε, και άλλη πινακίδα. Μπορούμε αμέσω να δούμε μέσω του, τσίπ αυτού εάν ε, είναι κλεμμένο το αυτοκίνητο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, μπορούν να κάνουν τέτοιου ελέγχου στα καναδικά σύνορα, πιν. Δεν είναι ακριβό. Αν αυτο, ο κάθε ε, οδηγός πληρώνει λιγότερο από ένα ευρώ για αυτό το σύστημα. Κάτι άλλο τώρα. Πρέπει να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση της αξιοπιστίας μας, της αξιοπιστίας του αυτοκινήτου, του κταίου δηλαδή. Αν εσύ έχεις ελέγξει το αυτοκίνητό σου στη Γερμανία, ε, κανονικά, και μετά αλλάξεις χώρα, ε, πρέπει να ξαναπεράσει κταίω στη νέα χώρα. Αυτό είναι περιττό, είναι επικάλυψη. Θέλουμε να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση αυτών των δοκιμών, αυτών των τεστ σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και αν πά, ας πούμε, ε, στην, αν πάει κανείς στην Ισπανία για τρεις μήνες για να σπάσει λίγο το χειμώνα και τη μαυρίλα του, δεν έχει κανένα νόημα να ξαναπεράσει αυτό το τεστ. ανοίγει κάποιο τη βάση δεδομένων, βλέπει ο αρμόδιος ότι έχει ε, περάσει κταίο σε μια χώρα και ισχύει αυτό για όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η επισκόπηση. Έχω ήδη το χρονοδιάγραμμά μου εγώ έτοιμο, αλλά καλό είναι να ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές για να δω τι άποψη έχουν για τις προτάσεις μου και αν πιστεύουν ότι βελτιώνουν την πρόταση της Κομισιόν, θα ήταν καλό αυτό. Ο κύριος Κάρας. Με ρώτησε τι κάνω με τις επαγγελματικές πινακίδες. Να μου πούνε στην άλλη, τι νομίζουν. Good. Right. Well, let's hear from the shadows. Yeah, professional vehicle registrations are included in the... Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε πρώτα τον ε, κύριο Κάρας και ότι συγγετή μετά την κυρία Στάιλερ, Ρίουλερ και τον υποφαινόμενο στο τέλος κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντερς, τον εισηγητή για την εξαιρετική προεργασία για τον φάκελο αυτό. Με την έκθεση αυτή διατυπώνουμε μία από τις κεντρικότερες ε, ανησυχίες που απασχολούν τους καταναλωτές αυτή την ε, εποχή αυτό το πρόβλημα ανήκει στα 22 σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που απασχολούν τους καταναλωτές και πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την διαδικασία έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη ενιαία αγορά. Τώρα δεν θα αναφερθώ σε κάθε ένα από τα σημεία. Να πω ότι Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην διαδικασία μεταφορά ενό αυτοκινήτου και σε περίπτωση άρνησης ε, της ε, μεταφοράς ε, ενός οχήματος από τη μία χώρα στην άλλη. Χρειαζόμαστε μια σίγουρη τράπεζα δεδομών, τραπεζα όπως η Γιούκαρης για παράδειγμα, όπως είπατε, και πρέπει να φροντίσουμε να καλυφθούν όλα τα κενά, να αποτρέψουμε την απάτη, την φοροδιαφυγή, να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη μας. Επίσης, σε περιπτώσεις σε καταχώρησης που δεν είναι εμπρόθεσμες, ε, θεωρώ πως πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, να προβλέπονται κυρώσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που είναι τώρα έξι μήνες για την καταχώρηση ενός ε, οχήματος. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να αλλάξει. Υπάρχουν προτάσει και για μικρότερο χρονικό διάστημα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίση, η αιτιολόγηση τη άρνηση χορήγηση σε μια τέτοια αδείας καταχώρηση πρέπει να είναι σαφής. Διότι φυσικά έχουμε να κάνουμε πέραν όλων των άλλων και με την ασφάλεια στους δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι σωστά και εγκαίρος και εμπρόθεσμα καταχωρημένο ένα όχημα. Αυτά προς το παρόν από εμένα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά μέχρι τώρα. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας και τους υπόλοιπου και οδησηγητέ. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση τη Επιτροπής και το στόχο της που είναι απλό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης. Αυτό είναι και ευχριστό για τους οδηγούς, αλλά και πολεμά το διασυνοριακό, τις διασυνοριακές, διασυνοριακές παράνομες δραστηριότητες ό,τι αφορά φαλκίδευση, κλεμμένες πινακίδες και το καθεξής. Τώρα, για τις διατυπώσεις ταξινόμησης, άρθρο 4.1. Το είπε και ο κύριος Μάντερς προηγουμένως. Σε ορισμένες χώρες ε, ε, ε, είναι το θέμα των πινακίδων αρκετά ευαίσθητο. Ε, στη σκοτία τουλάχιστον σίγουρα είναι. Είναι αρκετά σαφές το άρθρο 4.1 και η εξάμεινη περίοδος είναι υπερβολικά εκτεταμένη. Να μπορούμε να έχουμε άμεση ταξινόμηση για μόνιμες μεταφορές και μεγάλες περιόδους χωρίς ταξινόμηση δημιουργούν μια έλλειψη ασφάλειας και ασάφεια. Ενώ αν έχουμε σε συντομότερες μεταβατικές περιόδους θα έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια και θα περιορίσουμε και τους έμεσους φόρους κατανάλωσης. Δεν θέλουμε έμεσα η οδηγία αυτή να ενισχύσει την φοροδιαφυγή. Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει και προϋποθέσεις για την ταξινόμηση, με ανησυχεί το εύρος των ε, πληροφοριών που απαιτούνται ε, δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό ο αριθμό των πληροφοριών που ζητάμε. Μην ξεχνάτε ότι η οδηγία αυτή στόχο και την απλούστευση των διατυπώσεων και των διαδικασιών για του πολίτε. Σε πολλέ χώρε, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται και η ασφάλιση του αυτοκινήτου ω προπόθεση για την ταξινόμησή του. Ε, κάτι τέτοιο όμω ίσω επηρεάσει αρνητικά τι προσπάθειε ε, ε, τη καταπολέμηση ε, τη οδήγηση χωρί ε, κάλυψη από ασφάλεια. Θέλουμε υψηλό επίπεδο δικής ασφάλειας και σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση για τις φυνακίδες, όπως ξέρετε, προτιμούμε να κρατήσουν τα κρατημέρια της δικής τους άδειε για τις πινακίδες και ε, ιδιαίτερα τόνισα ε, το σκοτσέζικο πρόβλημα. Θέλουμε να κρατήσουμε τις δικές μας πινακίδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρήση της ραδιοσυχνότητας για να περιοριστεί ο αριθμός των παράνομων ε, κυκλοφορία πινακίδων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο μηχανισμό να χρησιμοποιηθεί και είμαι υπέρ τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και συμφωνώ με την πρόταση για τα αλλαγή των πληροφοριών με τη χρήση του φυστάμενου συστήματο ΕΟΚΑΡΙ. Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Αυτό είναι το ζητούμενο και κοινό μα στόχο. Ευχαριστούμε κύριε Μάντερ για την έκθεση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και περιμένω με ανυπομονησία τις συμβαστικές τροπολογίες και λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή, διότι πραγματικά συμπεριέλαβε όλα αυτά που ήθελα και εγώ να πω και το ζήτημα της ασφάλειας, όπως ανεφέρατε και, εσεί, κυρία Στάιλερ. Και τις ε, περιβαλλοντικές ζώνες Δηλαδή πραγματικά η έκθεσή σας τα έχει όλα. Πράγματα που δεν είχε ακόμα ούτε καν η Κομισιόν. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα με την βάση ε, Ουκάρης. Βρίσκω πάρα πολύ καλή την πρότασή σα. σω όμω θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ε, εξηγήσει, να μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε. Σε γενικέ γραμμέ είναι πάρα πολύ καλή έκθεση και χαίρομαι πολύ για την επόμενη συνεργασία μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω για τις πινακίδες, κύριε Μάντες, Η απάντησή σας ήταν έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Πιστεύω πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόοδο σε αυτό το θέμα με τις πινακίδες, διότι Επί του παρόντος ε, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια για τους ε, πολίτες. Όμως ε, έχω ορισμένες σκέψεις σχετικά με τις προτάσεις του κύριου Μάντες. Ναι, μεν πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα, όμως αυτό εξαρτάται και από τις ικανότητες των κρατών μελών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το σκεπτικό ότι αυτό είναι πρόδρομος της εισαγωγή ενός πανευρωπαϊκού συστήματος καταχώρησης αυτοκινήτων, βάσει δεδομένων δηλαδή, είναι πιστεύω τελείως αντιπαραγωγικό αν θέλουμε να είμαστε γρήγοροι. Και πράγματα όπως οι πινακίδες και απαιτήσει για έκδοση πινακίδων και το τσιπάκι με την ταυτότητα είναι πάρα πολύ ωραία, εφάνταστα, χρήσιμα, εμπλουτίζουν και διανθίζουν μια έκθεση, αλλά ειλικρινά αυτό που πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα απολύτως αναγκαία που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές και θα εφαρμόσουν το σύστημα το γρηγορότερο δυνατόν, διότι πιστεύω πως καταρχάς πρέπει να πούμε στην ε, Επιτροπή, της οποίας η πρόταση μου φαίνεται καλή. Να πω ότι η πρότασή σας είναι κάπως ακατάλληλη όσον αφορά την εισαγωγή ενός κοινού τύπου ταξινόμησης οχημάτων. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε αυτό το κοινό ενιαίο σύστημα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τα επιμέρους συστήματα να επικοινωνούν καλά μεταξύ τους και να συνδέονται με καλό τρόπο. Ωραία αυτά που μας λέτε, πολλές πληροφορίες, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσατε να οργανώσετε μία ακρόαση, γιατί πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ε, έχουμε ακούσει εδώ και θα μας ενδιαφέρε πιστεύω να μάθουμε περισσότερα. Αυτό που πρέπει να δώσουμε, σε αυτό που πρέπει να δώσουμε βάση είναι η ανταλλαγή δεδομένων και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το θέλουμε γρήγορα και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε τι, τι να κάνουμε. Ας πάρουμε αυτά που έχουμε τώρα, ας τα βελτιώσουμε και ας κάνουμε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να τα εφαρμόζουν. Και αυτό με τη σειρά του θα επιφέρει βελτιώσεις και σε άλλους τομείς. Και αυτό θα συνάδει και με τις ε, άλλες ενέργειες που κάνουμε ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, τους ε, τεχνικούς ελέγχους των ε, οχημάτων. Έχουμε προτείνει μία έκθεση για αμοιβαία αναγνώριση του τεχνικού ελέγχου, των ΚΤΕΟ. Και πραγματικά ε, ε, θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρημα... Επιχειρήσεων ότι είναι πολύ καλό, θεωρώ, πως ε, θίξατε και εσείς αυτό το θέμα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Είναι ένα κεντρικό σημείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χρειάζεσαι να περνά το όχημά σου αποκτέω σε κάθε χώρα. Αλλά πρέπει να δούμε τι είσαι προδιαγραφές για αυτούς τους τεχνικούς ελέγχους. Πρέπει να υπάρχουν κοινέ προϋποθέσεις και η πρόταση της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης MOVE πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις ε, δικές μας και με, την με, τις δικές μας προτάσεις. Η δική σας συνεισφορά που βρήκα αρκετά χρήσιμη είναι η καταγραφή των χιλιόμετρων που διανύει ένα όχημα. Και πιστεύω ότι ένας απλός έλεγχος απλά των χιλιόμετρων που έχει γράψει ένα αυτοκίνητο στο σύστημα ταξινόμησης θα αποδείξει εάν κάποιος αγοράζει αυτοκίνητα σε μία χώρα φτηνά και τα, πουλά σε, τα μεταφέρει σε μια άλλη χώρα και τα πουλά για να βγάλει κέρδος. Πιστεύω πως αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι πάρα πολύ απλό να το δούμε. Εγκρίνω λοιπόν την πρόταση Μάντερς προσωπικά. Διότι αυτό που θέλω είναι να μην δώσω, να δώσω όσο το δυνατόν λιγότερες ε, αφορμές στα κράτη-μέλη για να φέρουν αντιρρήσεις στην εφαρμογή του συστήματος. Δικό σας έργο, κύριε Ισηγητά, είναι να φροντίσετε αυτό να γίνει γρήγορα, αλλά παρακαλώ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εισαγωγή νέων συναρπαστικών μεν, αλλά πολύ δύσκολων δε απαιτήσεων. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μιλήσει. Κυρία Πέλτς, θα έρθει η σειρά σας σύντομα, αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες, ε, γιατί θα προετοιμάσω την γνωμοδότησή μου. Δεν φτάσαμε ακόμη στο δικό σας θέμα, κυρία Πέλτς. Okay. Um, I was going to... Σε λίγο, σε λίγο θα σας δώσω το λόγο. Ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκόγκα από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα παρέλθω στον εισηγητή μας, τον κύριο Μάντερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Μάντερς για την έκθεσή του. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεσή σας και υποστηρίζει και οποιαδήποτε βελτίωση ή εμπλωτισμό της έκθεσης της, της πρώτης επιτροπής προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να καταπολεμηθεί το έγκλημα ή παράνομε δραστηριότητε σε σχέση με τα ξυνόμιση και τι πινακίδε. Άλλωστε, απότερο σκοπό μα είναι η απλούστευση τη καθημερινότητα και τη ζωή των ε, πολιτών. Και χαίρομαι που με την έκθεσή σα ε, εστερνίζεστε το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βασικός κανόνας της πρότασης προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη δίνονται να ζητήσουν επαναταξινόμηση του οχήματο αν ο κάτοχος της πινακίδας έχει την κανονική του μόνη κατοικία στο κράτος αυτό. Και αυτή είναι η βασική αρχή της έκθεσης. Ελάχιστες αλλαγές υπάρχουν στο άρθρο 3. Δεν έχουμε αντίρρηση και χαίρομαι πάντως που η βασική αρχή της πρότασης παραμένει μετάβλητη με τη μορφή που την κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, κάποια άλλα θέματα ίσονος σημασίας που είναι απαραίτητο όμως χάρη συνέπεια και συνάφειας. Καταρχήν, ε, ορισμός του κατόχου του πιστοποιητικού ταξινόμησης. Είναι ένα θέμα που συναντάται και σε άλλα νομοθετήματα, την οδηγία 937 για παράδειγμα. Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή του ορισμού του κατόχου πιστοποιητικού ταξινόμησης ε, να γίνεται ταυτόχρονα και στην τελευταία πρόταση και στις προηγούμενες, γιατί αυτή είναι νέα πρόταση και καλό θα ήταν υπάρχει ευθυγράμμιση των διαφορών νομοθετικών προτάσεων. Εμείς προτιμούμε τον ορισμό όπως τον έχουμε υποβάλει, χωρίς αλλαγές. Και υπάρχει και ένα θέμα με το φόρο, με τη φορολογία. Εμείς ε, δεχθούμε οτιδήποτε αποτρέπει την ε, διάπραξη κλιμάτων ή την ε, χρήση πλαστών πινακίδων ή τις λαθροχειρίες σε τέτοια θέματα, αλλά αυτά μπορούμε να τα έχουμε μόνο για μεταχειρισμένα ή επαναταξινομημένα αυτοκίνητα αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο να την επεκτείνουμε σε όλα τα οχήματα και στην πρώτη ταξινόμηση και όχι μόνο στην επαναταξινόμηση, γιατί προς το παρόν η πρόταση περιορίζεται στην επαναταξινόμηση και όχι στην πρώτη ταξινόμηση του, εγγράφου, του οχήματος. Σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Και εδώ περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων. Ίσως απαιτηθεί τέτοια προϋπόθεση. Κάποιες χώρες ήδη το προβλέπουν και ίσως μια γενίκευση έχει νόημα. Και γενικώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει τη συνέχιση των συζητήσεων για να δούμε πώς θα διεξαχθεί και περαιτέρω η συνεργασία μας και η συζήτηση. Κύριε Μάντες, για να ολοκληρώσετε. Uh, uh, ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ για την υποστήριξη τα περισσότερα. Η ασφάλεια είναι μέσα, τα χιλιόμετρα είναι μέσα, στο παράδειγμα ένα. Για τη βάση δεδομένων, τι θέλω να βάλω, τον κοινό μορφότυπο της ταξινόμησης, ούτως ώστε να είναι αναγνώσιμος και αναγνωρίσιμος σε όλη την Ευρώπη. Σαν διαβατήριο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο ορισμός του κατόχου. Κάνα πρόβλημα δεν έχω. Ήμουνα... Υπάρχει και ακρόαση του Ιουνίου που έθεσε το εξής ερώτημα ή μάλλον η μαλλον η κρόση που κάναμε ε, έθεσε ε, το εξή ερώτημα. Ε, στο όνομα ποιανού θα είναι, στο όνομα του ατόμου ή στο όνομα της εταιρεία του. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Και εγώ γι' αυτό λέω να το κρατήσουμε όπως την οδηγία 99-77. Χαίρομαι σας που λέτε ότι σας αρέσει το κείμενο, αλλά για το θέμα της επαναταξινόμησης Καλό θα ήταν να αντιγράψετε αυτό που λέτε εδώ και σε άλλους σχετικούς κανονισμούς. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τεχνικές που έχουμε στην παλέτα μας για να αποφύγουμε την απάτη και να διευκολύνουμε την ε, ζωή όλων. Ε, επίσης, ο αριθμός πινακίδων. Δεν ζητάω κοινό αριθμό πινακίδων. Ο εθνικός κώδικας ε, ρυθμίζεται από διάφορες νομοθεσίες. Επομένως, ε, βασικά ε, τα αρχικά για τη χώρα είναι σαφή, απλώς η ιδέα είναι ότι ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει χρώμα άλλης χώρας. Σε 6 Ιουνίου είναι η ημερομηνία για τις προθεσμίες. Παρακαλώ συναδέλφους να μου στείλουν να λιγότερες ε, τροπολογίες. 27 Ιουνίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και να δούμε αν μπορούμε να συμβαστούμε τον Ιούλιο, γιατί θέλουμε να ψηφίσουμε στις 9 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω κάτι και να με βοηθήσει η Κομισιόν. Μιλήσατε για, το μορφότυπο. Υπάρχει κοινό μορφότυπος ε, στα έγγραφα ταξινόμησης. Υπάρχει, έτσι δεν είναι. Δεν ακούσαμε την απάντηση. Υπάρχει, αλλά δεν χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη-μέλη, μάλλον, είπε ο κύριος Μάντερς. Υπάρχουν κάποια θεματάκια γύρω από εκεί. Υποχρεωτική ασφάλιση, η μορφή της ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Από ό,τι ξέρω όμως, δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις. Επίσης, το Ιουκάρις Έξι κράτη-μέλη συμμετέχουν, αλλά τώρα είμαστε 28 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ήθελα την, ε, να επεκτείνουμε το Ιουκάρι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο, ο μορφότυπος του πιστοποιητικού ταξινόμησης ε, έχει προσδιοριστεί από την οδηγία 9937. Έχει υποχρεωτικά στοιχεία και προαιρετικά στοιχεία. Δηλαδή, κάποια κράτη-μέλη μπορεί να μην ε, συμπληρώσουν κάποια πράγματα. Τα υποχρεωτικά βέβαια πρέπει να υπάρχουν παντού στα πιστοποιητικά, αλλά υπάρχουν και τα προαιρετικά που ένα κατασμό μπορεί να επιλέξει να μην τα συμπληρώσει. Εσεί λέτε λοιπόν, λέτε να επεκτείνουμε τα υποχρεωτικά στοιχεία. In our proposal, we are based... Στην πρότασή σα, αυτό λέτε. Όχι, εμεί στην πρότασή μα ακολουθούμε αυτά που γίνονται στην οδηγία. Δηλαδή, αν αλλάξει 9937, τότε θα κάνουμε τι ίδιε αλλαγέ και εδώ. Θα είμαστε σε επαφή και θα τα συζητήσουμε αυτά. Γιατί αν υπάρχει ήδη κανένα πρόβλημα. Αλλά μια και κάποια στοιχεία είναι υποχρεωτικά και κάποια άλλα είναι θελοντικά, υπάρχουν διαφορές. Uh, Τότε η οργάνωση γερμανική μου είπε να βάλω αυτό το στοιχείο. Παρακαλώ, καλό είναι να επικεντρωθούμε στο τρέχον σύστημα, να μην ε, το αλλάζουμε για να μπορέσει να περάσει γρήγορα το κείμενο. Ποιο θα φανταζόταν θα είσαστε τόσο ζωντανή πέμπτη απόγευμα. Δεν θα το φανταζόμουν. Ε. Σα ευχαριστώ γι' αυτό. Και τώρα έχουμε να ακούσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Η κυρία Ιντικό Γκαλπέλτ που περιμένει. Η κυρία Ριούλε και εγώ είμαστε οι μόνοι σκιώδει συζητητές. Εγώ βέβαια δεν είμαι επίσημο ε, σκιώδει συζητητή, αλλά καλύπτω κάποιον άλλο. Πού είμαστε στη συζήτηση του προπολογισμού, κυρία Γκαλπέλτς. Έχουμε και ουγγρική μετάφραση. Τώρα μπαίνω στην καμπίνα η Διερμηνής. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε τη γλώσσα σας. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την δυνατότητα που μου δίνετε να σα παρουσιάσω τα πιλωτικά προγράμματα και τα το προπαρασκευαστικό έργο σε σχέση σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό του 2014. Okay. Okay. I, I start again. <laughs> okay. Okay. Okay. Thank. Αρχίζω από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω, όπως είπα, το πιλωτικά προγράμματα και τα προπαρασκευαστικά μέτρα σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό του 2014. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πιλωτικά προγράμματα, με προπαρασκευαστικά μέτρα για τον προϋπολογισμό του 2014. Προφανώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα τη διαμηνία, λέει ο προεδρος χρειαζομαστε Χρειαζόμαστε ένα-δύο λεπτά μέχρι να συνδεθούν όλοι οι διερμηνεί για να σας ακούσει όλος ο κόσμος στο ίντερνετ. Θα προτιμούσατε ίσως να περιμένετε δύο λεπτά και να έχετε κοινό δισεκατομμυρίων. Nobody else from the S&D is here shadowing the budget. So... Κανείς από τους σοσιαλιστές δεν είναι εδώ, σκιώδης ηγητής για τον προπολογισμό, οπότε αν θέλετε ευχαρίστω τον αναλαμβάνετε. You had a wastage, but anyway, I mean, we did our best, but we, we did shuffle around. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πρέπει όμως να μιλήσετε με την ομάδα σας, γιατί και ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ φαίνεται πως ξέχασε κάποια πράγματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Right, okay. Um, is it in English? Or? No, no, in English it's two. It's, Okay, no all right. For you. Okay. No chance for you. So Hungarian's on channel 14, if you want them to listen to in way of somebody for interpretation. But otherwise we're ready to go. Έτοιμοι είμαστε λοιπόν. Κυρία Γκάλ αρχίστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Παρότι δεν έχουμε πολλούς παρευρισκόμενους, ε, ενδεχομένως είναι πάρα πολύ αργά και έχουν φύγει όλοι, πάντως είναι ανοιχτά τα ερωτήματα που αφορά τώρα το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ μπορώ να σας πληροφορήσω για τις προτάσεις μου που είναι στα πλαίσια του προπολογισμού 2014. Έχει να κάνει με προπαρασκευαστικά μέτρα και ορισμένα πιλωτικά προγράμματα. προτάσεις μου έχουν διαβιβαστεί σε εσάς, τους ευρωβουλευτές, σε έντυπη μορφή, στην κυρία Ρούλε. Έχω λοιπόν ένα φυλάδιο που έχω συνοψίσει τις προτάσεις μου. Καταρχάς, το φόρουμ της ενιαίας αγοράς είναι ένα προπαρασκευαστικό μέτρο και πιστεύω ότι είναι κάτι σχετικά ε, εύκολα να κατανοήσουμε. Αυτό το φόρουμ είναι κάτι στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Το φόρουμ αυτό μπορεί να διοργανωθεί από το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα φόρουμ που αφορά την ενιαία αγορά και φυσικά αυτό το φόρουμ είναι κάτι που θα χρειάζεται συνεχή χρηματοδότηση. Προτείνω λοιπόν Επειδή ακριβώ αυτό το φόρουμ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φέρει κοντά τους καταναλωτέ, τους οργανισμού καταναλωτών, τα κράτη-μέλη τους, αντιπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να του ε, συγκεντρώσει λοιπόν μαζί και να του ε, δεσμεύσει να εφαρμόσουν την ε, νομοθεσία που αφορά την έννοια ε, αγορά. 2013 λοιπόν, το ποσό που προβλέπεται είναι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το φόρουμ. Αυτό το φόρουμ, όπως είπα, πρέπει να έχει συνεχή χρηματοδότηση. Η ενιαία αγορά είναι πλέον 20 χρονών. Και αυτό αφορά 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Είναι εξαιρετικής σημασίας. Έχουμε Πολλέ δυνατότητες που έχουν μείνει ακόμα ανεκμετάλλευτες. Έχει δημιουργηθεί μια έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πολλές φορές αναφέρουν ότι υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, προβλήματα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τις ε, διακρίσεις ε, στις συνθήκες απασχόλησης και τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την διαδικασία ε, προκηρύξεων για δημόσιες προμήθειες. Αυτό προσδιορίζεται συνήθως ε, σε έλλειψη πληροφόρηση, σε μη τήρηση των κανόνων και σε ορισμένες φορές ε, σε έλλειψη των κανόνων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο φόρουμ, έτσι οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να έχουν άμεση συμμετοχή και να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να επηρεάσουν λοιπόν έτσι την λειτουργία της ενίας αγοράς. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολιτικά σημαντικό να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά διαστήματα τις ε, λειτουργίες του. Θα πρέπει να δημοσιεύονται τακτικές ε, εκθέσεις, ε, για παράδειγμα στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, να υπάρχουν εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα κοινοποιούνται τακτικά. Φυσικά, είναι γνωστό τη πάση ότι οι καταναλωτές πολλές φορές έχουν έλλειψη πληροφοριών, δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους και πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το φόρουμ θα μπορέσει να είναι μια πηγή πληροφοριών αυτών. Να αυτά για την πρώτη πρόταση, να περάσω τώρα στην δεύτερη μου πρόταση, το YET, το Your Europe Travel. Είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ξέρετε όλοι λοιπόν τα apps στα, στα κινητά. Η πρότασή μου λοιπόν έχει ως εξή τα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μια εφαρμογή για κινητά, η Ευρώπη για σας, η δική σας Ευρώπη, μια πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Πολλέ φορέ λοιπόν, όταν οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν δυσκολίε, είτε αυτέ είναι όταν θέλουν να ψωνίσουν κάτι σε ένα κατάστημα ή όταν πάνε διακοπέ. Έχουν προβλήματα λοιπόν με την γλώσσα, με το σύστημα και γι' αυτό λοιπόν αυτή η εφαρμογή θα, μπορούσε, θα μπορεί να τους παρέχει ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Εδώ να πω ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν λάβει πολλά μέτρα, έχουν κάνει πολλά βήματα για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αυτό όμω δεν ισχύει παντού σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχει γίνει μια μελέτη η οποία διαπιστώνει ότι ο αριθμός των χρηστών ε, smartphone, έξυπνων κινητών τηλεφώνων έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν εκπλήσει κανέναν φυσικά. Και είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι στο μέλλον ο Λεώνα και περισσότεροι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν smartphone, τα ξυπνά κινητά τηλέφωνα. Και λοιπόν η εφαρμογή αυτή θα μπορεί να σταθεί να βοηθήσει πάρα πολλού. Για παράδειγμα, είσαι σε ένα αεροδρόμιο, ακυρώνεται η πτήση σου. Με την εφαρμογή αυτή θα μπορεί να ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται με την πτήση σου και τα δικαιώματά σου αν είσαι επιβάτης, πώς μπορείς να ασκήσεις λοιπόν και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου και όλα αυτά από το κινητό σου τηλέφωνο. Αυτό επίσης δεν περιορίζεται μόνο στο, στα αεροπορικά ταξίδια αλλά και στις αγορές και στα εμπορικά καταστήματα. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι, να διατυπώσω ένα ερώτημα, να πω ότι στην πρότασή μου δεν αναφέρομαι σε αυτό. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στην ε, επαλήθευση του προγράμματος αυτού. Υπήρξαν κάποια προβλήματα με την χρηματοδότηση και τα ε, όργανα τα οποία τα χρηματοδοτικά όργανα. Η κυρία Ρούλε ε, έχει ασχοληθεί με αυτό. Αναφέρομαι στην ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Υπάρχει ένα σχέδιο έκθεση στο οποίο αναφέρεται η εναλλακτική λοιπόν επίλυση διαφορών. Ο στόχος είναι να προωθήσουμε αυτή την εναλλακτική επίλυση διαφορών ανάμεσα στους καταναλωτές και στους παρόχους υπηρεσιών σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών. Να πλουστεύσουμε λοιπόν την διαδικασία αυτή. Τώρα η προθεσμία για την ε, εφαρμογή είναι το 2015 της επίλυσης διαφορών. Όμως η εμπειρία μου δείχνει ότι πρώτα πρέπει να διεξάγουμε εκτενέστατες δοκιμές με τους καταναλωτές έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους ένα σύστημα επίλυσης διαφορών που να λειτουργεί. Οι συνάδελφοί μου έχουν επικοινωνήσει ήδη με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά υπάρχει μια ε, στήριξη της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης στην πρότασή μας. Η χρηματοδότηση όμως είναι ένα πρόβλημα. Η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του προγράμματος προστασίας των καταναλωτών. Στις επιλύσεις διαφορών σημαντικό είναι όλα τα ένδικα μέσα να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Όμως το πρόβλημα με την ε, μετάφραση εδώ είναι οικονομικό. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια γι' αυτό. Θα μπορούσαμε ίσως να μετατοπίσουμε κονδύλια, για παράδειγμα, από, την, ε, από το Connecting Europe, από το Συνδέοντας την Ευρώπη. Όμως αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο. Είναι ένα θέμα που μας καίει για τα κονδύλια. Εάν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα κονδύλια που θα διατίθενται στα πλαίσια του προϋπολογισμού, αυτό θα ήταν φυσικά ευκταίο. Είμαι ανοιχτή όμως, μια και το ερώτημα είναι αρκετά επίμαχο, σε προτάσεις και σε σχόλια των υπολείπων. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την τρέχουσα κατάσταση του προϋπολογισμού. Χθες δεν καταφέραμε να έχουμε περισσότερε και νεότερε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, να σα πω ότι δεν γνωρίζω τα μέσα και τα έξω των διαδικασιών του προπολογισμού. Να σα πω όμω ότι πρέπει να μα παρουσιαστεί κανονικά μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Οι προθεσμίε δεν έχουν αλλάξει και στην πρότασή μου θα μπορούσα να ενσωματώσω τις προσωπικές μου εμπειρίες μέχρι τώρα. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω αυτή την παρουσίαση και με χαρά μου θα ακούσω τις ε, αντιδράσεις και τα σχόλιά σας. Uh, good. Well, thank Thank ευχαριστούμε κυρία Πέλτ. Συζητήσαμε το θέμα του προϋπολογισμού χθες ε, για την ε, επιγραμμική επίλυση διαφορών Solvit. Και ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό του προπολογισμού και αναφέρθηκε στην πιθανότητα να βγουν τα κονδύλια από άλλες γραμμές. Αλλά εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για το Connecting Europe και δεν ξέρω, α, δεν μπορούμε καν να υποβάλουμε σχετικές συστάσεις. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Ρούλε να σχολιάσει. Ναι, πολύ σύντομα σχόλια. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια, διότι το έργο τη ήταν δύσκολο. Δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα τι διαπραγματεύσεις και δεν γνωρίζετε πλήρως την γραμμή του προπολογισμού και πραγματικά ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις προτάσεις σα Φυσικά για εμά. είναι δύσκολο να κάνουμε πράγματα εφόσον δεν γνωρίζουμε και να δώσουμε πράσινο φως εφόσον δεν γνωρίζουμε τη γραμμή του προπολογισμού. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε και μετά να ενεργήσουμε πάρα πάρα πάρα πολύ γρήγορα όταν έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν τα σχέδια. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την προετοιμασία σας. να κάνω εγώ ένα σύντομο σχόλιο. Α, καλό θα ήταν αν μπορείτε να μας υποβάλλετε το εγγραφό σας για το ADR και τη θέση σας. Θα μας βοηθήσει χθε οι συντονιστές. Συμφωνήσαμε με τις γενικές κατηγορίες για τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα καταναλωτών αλλά θέλουμε συγκεκριμένε πληροφορίες για τα επιμέρους πιλωτικά προγράμματα. Τώρα για το δεύτερο θέμα, αυτή την ε, ταξιδιωτική εφαρμογή δεν είμαι ενήμερο, αλλά από ό,τι ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα εκδοχή της, του πακέτου οδηγιών, του, της για, το για τα ταξιδιωτικά πακέτα. Μια εξυγχρονισμένη εκδοχή που φυσικά θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με και η δική μας πρόταση με, την, με τις νέες νομοθετικές προτάσεις. Δεν έχει νόημα να προτρέξουμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτεραιότητες της δικής μας Επιτροπής, η πλατφόρμα για τις ε, online επιλύσεις διαφορών και το δεύτερο θέμα είναι ε, θέματα σημαντικά και ε, για το δεύτερο θέμα το ταξιδιωτικό, το Europe, Your Europe Travel και τη σχετική εφαρμογή δεν νομίζω ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα αλλά καλό θα ήταν αυτά να τα θέσουμε και στους συντονιστές για να δούμε ποια είναι η δική τους γνώμη. Θέλετε το λόγο πάλι για μια ανακεφαλαίωση, να συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας, συνάδελφοι. Σίγουρα αυτή η εφαρμογή Your Europe Travel, η Ευρώπη σας δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Δεν είμαστε σαφείς και σίγουρα θα μας βοηθήσει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα πρωτού ολοκληρώσουμε την πρόταση. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να συνατύχει πλήρους υποστήριξης. Σαφέστατα. Δεν όσο για το φόρουμ της ενέας αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί λοιπόν στην πρόταση. Θα σας παρακαλούσα να μην το πετάξουμε, να μην το παραμερίσουμε, να το κρατήσουμε εδώ στην ημερήσια διάταξη μέχρι να έχουμε νεότερα με τα ADR και να δούμε μετά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 10 του μήνα θα έχει μεταφραστεί η πρόταση και εδώ στην Επιτροπή η πρόταση θα παρουσιαστεί επίσημα στις 8 ε, και 9 Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν έναν ολόκληρο μήνα για να το κοιτάξουμε, για να το επεξεργαστούμε, να δούμε την, ε, πώς μπορούμε να τον ενσωματώσουμε στη γραμμή προϋπολογισμού και μετά στις 19 ε, Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις Ιουλίου, συγγνώμη, είναι προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά σας και ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να το παρουσιάσετε ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διατάξης σήμερα. Απλά θα ήθελα στο τέλος να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι μια ειδική συνεδρίαση την επόμενη Τρίτη για την ε, ακρόαση επιβεβαίωσης του υποψήφιου Επιτρόπου κύριο Μίμιτς από την Κροατία. Θα αρχίσουμε στις 9.30. Θα μεταδοθεί η ακρόαση από το διαδίκτυο. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 17 Ιουνίου, από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και Τρίτη 18 Ιουνίου, 9 το πρωί και μετά 3 το απόγευμα. Θα χαρώ να σας δω όλους εκεί λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Γεια σας.